Colleagues, I'm going to make a start. We have a packed agenda, so thank you again. Θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ και πάλι τους αδέλφους που ήρθαν στην ώρα τους. Πρέπει όλοι να κάνουμε όμως μεγαλύτερη προσπάθεια να φτάνουμε στην ώρα μας. Ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Hey colleagues, uh, the adoption of the agenda. Um... Λοιπόν, όπως έλεγα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ο Υπουργός ε, της ε, Αυστρίας θα μας μιλήσει για μια πρωτοβουλία της Αυστρίας ε, σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Την 5η στις 4 του μήνα, 3 το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Η κυρία Γιωχάννα Μικ Λάιτνερ θα είναι εδώ. Επίσης έχουμε την ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση. Αναβάλλεται για τις 11 Δεκεμβρίου το θέμα αυτό. Επίσης στο σημείο 18 θα συζητηθεί από τις 10.30 έω τι 11.30 και το 17 θα επακολουθήσει και δει από τι 11.30 τι 12.30. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται η τροποποιηθήσα ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχει διαδικαστικό ο κύριος Βόιτ. Θέλετε το λόγο για τη διαδικασία. Παρακαλώ, σας ακούμε. Äh, Στις 4 ε, Σεπτεμβρίου ε, έχω ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία θεμελιωδών ε, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Το υπέβαλα λοιπόν και ακούω τώρα ότι αποφάσισαν οι συντονιστές να μην το θέσουν στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να ρωτήσω αυτό συνηθίζεται γιατί με βάση το παράγραφο 133 του κανονισμού το κατέθεσα και θα έπρεπε τουλάχιστον στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συζητηθεί. Οχτώ βουλευτές συνελήφθησαν στην Ελλάδα κάτω από ποιες συνθήκες. Γι' αυτό κατέθεσα αυτή την πρόταση και δεν θέλω να ε, αγνοηθεί. Παρακαλώ να με ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για το σημείο αυτό, κύριε Βόιτ. Ήταν ε, στην ε, ημερήσια διάταξη των συντονιστών. Δεν υπήρξε αντίδραση από τις πολιτικές ομάδες, αλλά μπορούμε να το καταθέσουμε εκ νέου, να το ξανασυζητήσουμε και θα σας πω. Αλλά ήταν ε, στην συνέντευξη των συντονιστών. Δεν αντίδρασαν απλά οι πολιτικές ομάδες. Υπάρχει και άλλο αίτημα επί της διαδικασίας. Παρακαλώ. Ποιος είναι ο... Δεν βλέπω την καρτούλα. Yeah, please go ahead. Harald από την Αυστρία. Κύριε Πρόεδρε, δεν το δέχομαι με αυτή τη μορφή αυτό. Είναι θέμα το πώς αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κανονισμό του. Είναι θέμα ε, δημοκρατίας και πώς ε, αντιμετωπίζονται τα κοινοβουλευτικά θέματα. Η συνεδρίαση των συντονιστών πρέπει να προετοιμάζει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Όχι όμως να αποφαίνεται για το ποιες προτάσεις από ό,τι ακούμε ε, θα αγνοηθούν και ποιες όχι. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες του Κοινοβουλίου και όταν υποβάλλονται προτάσεις ψηφισμάτων από μένα ή από οποιονδήποτε άλλον συνάδελφο ε, δεν μπορούν αντικανονικά να παραμερίζονται από τους συντονιστές. Αυτή είναι μια παράδεκτη κατάσταση και ζητώ να πάρετε θέση και εσείς κύριε Πρόεδρε. Και βέβαια να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι νομότυπες ε, προτάσεις να αντιμετωπίζονται σωστά διότι θα πρέπει με δημοκρατικό τρόπο να διαμορφώνονται οι απόψεις. Δυστυχώ όμω πρέπει να το δεχθείτε. Επαναλαμβάνω ότι ήταν ε, σημείο τη μέση διάταξη των συντονιστών. Αντίδραση από τι πολιτικέ ομάδε δεν υπήρξε. Θα επανασυζητηθεί. Θα επανέλθω και θα σα ενημερώσω. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Περνάμε στο σημείο 2. Σε ό,τι αφορά τις γλώσσες, ε, δυστυχώς δεν παρέχει τη διερμηνία στα δανέζικα, στα λετωνικά και στα κροατικά. Στο δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις ε, συστάσεις των συντονιστών δυνάμει του, του κανόνα μάλλον 205, ε, του εσωτερικού κανονισμού Γιάν Άλμπρεχτ από τους Πρασίνους θα είναι εισηγητής ε, της γνωμοδότησης επί της έκθεσης της πρωτοβουλίας Επιτροπής Σύνδεσης, τάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις ότι έφερε τη συμφωνία TTIP. Ο Γερούν Λέναρ ε, από το ΕΛΚΑ ορίστηκε εισηγητή για την γνωμοδότηση στην έκθεση Ήτρε για την ε, θέσπιση προγράμματο για λύσεις διαλειτουργικότητα ε, για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες, το ISA2. Διαλειτουργικότητα ως τρόπο για τον για τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Παίρναμε τώρα στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Κατά πολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτησης βάρους των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 26 Νοεμβρίου έλαβε χώρο τρίτος τριμερής διάλογος. Ο Χουάν Φερνάντο, ο συντονιστής μας, θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίχθηκε αυτός ο τριμερής διάλογος. Ε, ο κύριος ε, Λόπεθ Αγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Θα σας ενημερώσω λοιπόν για τις ε, διαπραγματεύσεις. Είπατε ότι έγινε για την οδηγία αυτή ο τρίτος τριμερής διάλογος και μάλιστα στη διάρκεια της Συνόδου Λομέλειας του Στρασβούργου μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω πει και σε προηγούμενες περιπτώσεις ότι η Ιταλική Προεδρία εργάζεται σκληρά ε, και δείχνει προσιλωμένη ε, στο στόχο της, εξε, της ε, επίτευξης σημαντικής πρόοδου για τις συνολικές διαπραγματεύσεις επί του θέματος αυτού την προηγούμενη εβδομάδα κατέστησε σαφές ότι μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου υπάρχει συμφωνία για κάποια σημαντικά ζητήματα ενδεχομένως και αυτό ίσως μπορεί να σημάνει ότι θα έχουμε επιτοσή με αυτόν συμφωνία σύντομα σε ό,τι αφορά την έννοια του public official του δημόσιου αξιωματούχου περιλαμβάνει και τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε σχέση και με μια προηγούμενη οδηγία, την οδηγία του 95. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για τα δικήματα που τιμωρούνται και με κάποιες ποινές μέχρι και κάθριξης. Ε, αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά ε, έχουμε το θέμα των κατοφλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Τα κατώτατα αυτά όρια. Και είναι και η προσέγγιση της ε, πρότασης πρόστιμα οικονομικά σε ό,τι αφορά ζημίες στον προπολισμό της Ένωσης λόγω πλεονεκτημάτων που απέκτησε ο δράστης, ο παραβάτης. Θα πρέπει να ορίζουμε τα δικήματα που κολλάζονται με ποινές κάθυρξης και ποια είναι η ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια. Πέντε έτη συγκεκριμένα είναι το κατόφλι. Όμως το Συμβούλιο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να την παρακάμψει την προσέγγιση αυτή του κατοφλίου και να αφήνει έτσι ευρύτερα περιθώρια εκτίμησης για τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και τους νομοθέτες ε, ε, που καθορίζουν τις διτάξεις του εθνικού ποινικού δικαίου. Εκεί λοιπόν έχουμε πρόβλημα, διαφωνία. Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, ε, τη λύψης του, στο πεδίο εφαρμογή οδηγία αυτό το θέμα δεν το έχουμε ακόμη θίξει ε, στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου. Είναι σημαντικό στοιχείο και για εμά πρέπει να περιλαμβάνεται ω ίδιο πόρο για την κατάρτιση του προπολογισμού τη Ένωση, ο ΦΠΑ. Η Ιταλική Προεδρία προτίθεται να θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων που θα γίνει αύριο. Και οι υπουργοί έτσι θα ολοκληρώσουν ε, το έργο της Ιταλικής Προεδρίας. Αλλά εάν δεν εξευρεθεί λύση που να είναι βιώσιμη για εμάς, από πλευρά Συμβουλίου, σημαίνει ότι η σκητάλη περνάει στην επόμενη Προεδρία ή τη στη Λετωνική. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει κάποια δυνατότητα σε επίπεδο Συμβουλίου ίσως και σε σχέση με τους Υπουργούς Οικονομικών για να δουν κατά πόσον θα πλακούμε στο θέμα αυτό του ΦΠΑ ή όχι. Ελπίζω να υπάρξει ευελιξία από τα κράτη-μέλη για να συμφωνήσουμε επί της οδηγίας και να μπορέσουν να συνεχίσουν αποδοτικά οι διαπραγματεύσεις. Και πάλι στην επόμενη ολομέλεια του Στρασβούργου να έχουμε περιθώρια λιγμών. Ιδάλλως, ίσως αναλάβει η, Ιταλική, η συγγνώμη, Λετωνική Προεδρία το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Και το ίδιο θα κάνουμε και για τον ε, τριμερή διάλογο για το ξέπλυμα χρήματος. Ναι, την περασμένη εβδομάδα έγινε στο Στρασβούργο τριμερής διάλογος και θα γίνει και σε δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο άλλος ένας. Είναι αυτός ένας φάκελος που τον έχουμε μαζί με την Επιτροπή ΕΚΟΝ Άρα δύο εισηγητές είναι παρόντες. Το πρόβλημα είναι ότι το Κοινοβούλιο θέλει ένα δημόσιο μητρό για τους ε, τελικούς δικαιούχους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε η κοινωνία να ξεκαθαρίζει θέματα όχι μόνο ξεπλήματος, ε, ε, αλλά και θέματα φοροδιαφυγής και φόρο αποφυγής. Ε, ε, είδαμε, τα, είδαμε το σκάνδαλο στο Λουξεμβούργο. Ε, οπότε βλέπουμε πώς αλλάζουν τα δεδομένα προκειμένου περιφορολογικών θεμάτων και στο τελευταίο τριμερή η πρόταση του Συμβουλίου για τη μορφή που πρέπει να έχει ένα τέτοιο κεντρικό μητρό δεν έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο γιατί ήταν πολύ περιοριστική σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση του κοινού και η Κομισιόν προσπάθησε, ε, υποσχέθηκε να κάνει μια νέα προσπάθεια αναδιατύπωσης. Είδαμε ένα non-paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ακόμα δεν το συζητήσαμε με τους σκιώδεις και δεν είμαι βέβαιη αν αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στον επόμενο τριμερή. Εν τω μεταξύ, χθες κοινοποιήθηκε μια επιστολή των Υπουργών Οικονομικών Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και λέει ε, πει έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να προχωρήσουμε στο θέμα φόρο διαφυγής. Για παράδειγμα, η ενωσιακή νομοθεσία μπορεί να δει ορισμένα τρας και άλλες μη διαφανείς ε, επιχειρήσεις με οργανισμούς και άλλες δυνατότητες ούτως ώστε να εντοπίζονται οι ε, δικαιούχοι και να είναι υπόχρεοι ε, για αφορολόγηση. Δεν λέει ε, δημόσιο ή κοινό μητρό, αλλά λέει ότι ένα μητρό είναι χρήσιμο για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Και αυτό φωτίζει με διαφορετικό φως του τριμερεί που είχαμε μέχρι τώρα, γιατί μέχρι τώρα ισχυρίζεται το Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινό δημόσιο μητρό για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, γιατί αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομικής μας βάσης. Αν όμως οι υπουργοί τρει αυτοί, Ιταλία, οικονομικών Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας ισχυρίζονται ότι μπορεί να αλλάξει αυτό, θα έλεγα ότι η συζήτηση ε, παίρνει διαφορετικό δρόμο. Θα ήθελα λοιπόν το μήνυμα αυτό να ε, περάσει στο Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Δεν ξέρω αν ήρθε η Ρόζι Μπίντι και η συνάδελφή της εδώ. Είναι καθοδόν. Πόσο καθοδόν. Τώρα δηλαδή έρχονται, μπαίνουν στην αίθουσα. Ε, δεν θέλω να ε, καθυστερήσουμε. Λοιπόν, ξέρουμε πού είναι. Α, η Άννα Γκόμες. Θα καλύψει το χρόνο μέχρι να έρθουν. Έχεις το λόγο. Ναι, μετά από αυτά που είπε η Τζούντι Αργεντίνη θα ήθελα και εγώ να πω ότι διαπιστώσαμε ότι πράγματι ε, πολλοί επιχειρηματίες ε, στον τραπεζικό τομέα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με ένα δημόσιο ή κοινό μητρό των ε, δικαιούχων. Και ε, ε, γι' αυτό είναι περίεργο ότι κάποιες κυβερνήσεις γερμανική ανθίστατο τώρα, μάλιστα μας λέει η Τζούντιθ, ότι ο Υπουργός ο Γερμανός υπέγραψε την επιστολή Οπότε νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμείνει στην θέση που υπάρχει στην έκθεση και την οποία τα δύο μέλη μας ε, ε, περασπίστηκαν στον τριμερή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ ενδιαφέρον γιατί αφορά την Επιτροπή Έρευνας ε, ε, για εγκληματικές, εγκληματικές οργανώσεις και τη μαφία. Ε, χαιρετίζω την Ρόζη και τα μέλη που μετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Έρευνας. Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψε με αυτή την αντιπροσωπεία από την Ιταλική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Γνωρίζουμε όλοι ότι και εμείς είχαμε μια ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος στην Επιτροπή Κρίμα. Πολλά μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που παρευρίσκονται και σήμερα μετήχαν και τότε εκεί. Ολοκλήρωσε η ΚΡΙΜ το έργο της πριν από ένα χρόνο όπως ξέρουμε. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συμμετέχει πάρα πολύ ε, σε όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν και από την Ιταλική Επιτροπή Έρευνας για την Καταπολέμηση της Μαφίας Οπότε είναι πολύ σχετικό το έργο των επιτροπών μας. Πέρσι εγκρίναμε νέους κανόνες για την δίμευση και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε νέες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος, τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, το Eurojust, την Europol κλπ. Και επίσης έχουμε και μια συζήτηση που τώρα συνεχίζεται σχετικά με την νέα ε, στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Οπότε θα γίνονται πάρα πολύ εντατικέ συζητήσεις και είναι και πολύ σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή να ακούσουμε από εσά τι κάνετε στο δικό σας κοινοβούλιο και τις δικές σας τις ε, δομές. Ε, χωρίς άλλη καθυστέρηση θα σας δώσω το λόγο και στους συναδέλφους σας ίσως να πούν δύο λόγια και να παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας. Είστε πολύ γνωστοί και στην Ιταλία και στους συναδέλφους ε, εδώ στην ΛΥΜΠΕ ε, για το έργο σας. Ε, λοιπόν, περιμένουμε τις δηλώσεις σας και θα ακολουθήσει συζήτηση. Η Ρόζι Μπίντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που προσκαλέσατε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ιταλικού Κοινοβουλίου να έρθει και να παρουσιάσει το περιεχόμενο της έκθεσής μας για το οργανωμένο έγκλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή ε, ε Προεδρία Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ένωσης. Η Γερουσία επίσης ομόφωνα έκανε δεκτή την σχετική πρόταση και σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσουν και νομίζουμε ότι θα είναι ομόφωνη και αυτή η ψηφοφορία. Αυτός είναι λόγος ε, να χαίρομαι και να συγκινούμε ε, διότι από το 98 μέχρι το 99 ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή ήταν η πρώτη μου κοινοβουλευτική εμπειρία, πολύ ε, χρήσιμη, έμαθα πολλά και η παρουσία μου σήμερα σε αυτή την ε, διευρυνόμενη κοινότητα που ελπίζουμε να συνεχίσει να διευρύνεται μου δημιουργεί μεγάλη ικανοποίηση. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Έρευνας ε, για το φαινόμενο της μαφίας ε, και άλλων εγκληματικών αλλοδαπών μεταξύ άλλων οργανώσεων που είχα την τιμή τις οποίες είχα την ε, τιμή να προεδρεύω δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1997 και ολοκλήρωσε το έργο της πριν από ένα περίπου χρόνο. Σε κάθε νομοθετική θητεία ανανεώνεται και επί 15 χρόνια η Επιτροπή κατά της Μαφίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, προχωρούσε το έργο της. Εμείς Μπορούμε να αρχίζουμε έρευνες ε, όπου αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμά μας. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η Ιταλία έμαθε πάρα πολλά πράγματα για το οργανωμένο έγκλημα και είναι επίσης η χώρα εκείνη όπου η μαφία και άλλες εγκληματικές οργανώσεις ε, καταπολεμήθηκαν πάρα πολύ. Είμαστε επίσης και έθνος καταπολέμησης της μαφίας. Διότι έχουμε αποτελεσματικότατα εργαλεία για τη ζημία που προκλήθηκε ε, όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε να καταπολεμούμε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα γνωρίζοντας ότι δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό θα πρέπει να την καταπολεμούμε και με ε, εργαλεία που δεν γνωρίζουν σύνορα. Ολοκληρώσαμε το έργο μας ε, σεβόμενοι τις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Χάρτας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και ολοκληρώνουμε τα εργαλεία μας για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή, η οποία υπήρχε επί 15 χρόνια και ε, όταν, ε, σε, εποχές όπου ε, δεν γινόταν παραδεκτή η ύπαρξη της μαφίας, τώρα, χάρη στο έργο της, που οδήγησε σε νέα νομοθεσία και ήλεγχε την αποτελεσματικότητά της, είναι σημείο αναφοράς για θέματα μαφίας και για προτάσεις ρυθμιστικές και κανονιστικές για να ε, βελτιώνονται τα υφιστάμενα μέτρα. Η νομοθεσία που θεσπίσαμε στη χώρα μου γεννήθηκε στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Μαφίας. Ε, εξαιρετικό έργο επετέλεσε ο πιο λαλατόρε, ο οποίος ε, δολοφονήθηκε από τη μαφία στο Παλέρμο το 82 οι αρχές του ακόμα είναι ζωντανές και μας εμπνέουν. Κατά τον πρώτο χρόνο της Επιτροπής, της διεδικής μας θητείας, τον Νοέμβριο του 2013, θελήσαμε άμεσα αυτή τη διαδικασία ε, της μαφίας, θελήσαμε να τη βάλουμε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Και ε, έτσι κάναμε μια μελέτη και διεθνή για να δούμε όλα τα φαινόμενα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι η Επιτροπή μας ε, έπρεπε να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του, των υφιστάμενων νομικών κανόνων. Επίσης έπρεπε να υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις ούτως ώστε τις διεθνείς ε, ε, για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων να τις βελτιώσουμε και έτσι να συμβάλλουμε ε, σε ένα χώρο ε, κατά της μαφίας και να προωθήσουμε μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Πάλι πάνω στη βάση της αρχικής νομοθεσίας η Επιτροπή μας έχει το καθήκον να εξετάσει τις αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο ή στο σύστημα παραγωγής λόγω της ύπαρξης και δράσης της μαφίας. Βλέπουμε ποιες αρχές ε, θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις όπως η ιδιωτική οικονομία, ελεύθερος ανταγωνισμός και άλλες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή συνειδητοποιήσαμε αυτό που είπε και ο κύριος Γκαραβίνη, το οποίο ε, θα έρθει εντός ολίγου, ότι η Επιτροπή αυτή ε, είχε σαν στόχο να συντάξει μια έκθεση ε, επευκαιρία της, του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας κάναμε μία λεπτομερή προετοιμασία ε, ελέγχου, ε, παρακολούθησης κτλ. για να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η, ποιο είναι το επίπεδο της Ιταλικής και της Ευρωπαϊκής ε, κατάστασης όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ε, γενικότερα παράνομες δραστηριότητες αλλά υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση στον τρόπο της διαχείρισης της ροής των μεταναστευτικών ε, ρευμάτων, ε, της ε, πορνείας και σε, άλλες, σε άλλα επίπεδα εγκληματικών δραστηριοτήτων. αυτό το οποίο επομένως συνειδητοποιήσαμε μετά από όλη αυτή την έρευνα είναι ότι το θέμα της ε, εγκληματικής, ε, των εγκληματικών οργανώσεων και των οργανώσεων που σχετίζονται με τη μαφία δεν αφορά μόνο μία χώρα. Άρα δεν είναι μία χώρα υπεύθυνη για να το αντιμετωπίσει. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν χώρο ε, δικαστικής συνεργασίας κατά της μαφίας έτσι όπως ακριβώς αναφέρεται και στο καταστατικό της Επιτροπής μας, αλλά έτσι και όπως το έχουν ευχηθεί και, διάφοροι, και το επιθυμούν διάφοροι ε, ευρωπαϊκοί θεσμοί. Εμείς πιστεύουμε και θέλουμε η εγκληματική δραστηριότητα, το οργανωμένο έγκλημα, να που ρυθμίζει, αν θέλετε, και πολλές φορές ε, και την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η διεύρυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την μαφία είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να προδικάσει και το μέλλον μας. Η ίδια η Ευρώπη σε όλες, μέσα από όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις ε, συνειδητοποιεί ότι η μαφία αποτελεί ένα βάρος σε όλες τις δραστηριότητές μας. Επίσης, χρειάζεται να, ε, να εξετάσουμε εις βάθος την ε, παράνομη οικονομία και το πώς αυτή επηρεάζει το κάθε ΑΕΠ και να δούμε και ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να υπολογίσουμε το, το καρπό, αν θέλετε, των εγκληματικών ε, ε, δραστηριοτήτων που είναι 126 δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 1% του ε, ευρωπαϊκού ΑΕΠ και 3,6% του εθνικού ΑΕΠ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το, το καρπό το αποτέλεσμα των εγκληματικών δραστηριοτήτων στο κάθε ΑΕΠ. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα πρέπει να εντείνουμε την, τον πόλεμο κατά των, αυτών των δραστηριοτήτων, διότι εμείς θέλουμε να έχουμε έναν πλούτο διάφανο, καθαρό. είναι πολύ ισχυρή η αρνητικό, αρνητικό, είναι πολύ ισχυρός ο αρνητικός πλούτος ο οποίος κυκλοφορεί στις οικονομίες μας. Και εμείς θέλουμε μια οικονομία που είναι ε, στην υπηρεσία όλων των πολιτών της ε, Ευρωπαϊκής ε, Υπήρου. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευαισθησία, μια κουλτούρα κατά της μαφίας στην Ευρώπη. Και όχι μόνο ε, στις χώρες που είναι εγκατεστημένες τέτοιες ε, εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και στις χώρες όπου διευρύνονται οι μαφιόζικες δραστηριότητες, διότι η μαφία δεν υφίσταται μόνο στην Ιταλία και η μαφία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από το γεγονός ότι οι ε, δραστηριότητες της μπορούν να ενταχθούν σε, διάφορα, σε διάφορες μάρκες που είναι γνωστές. Ε, η εισαγγελία κατά της μαφίας στην Ρώμη μπόρεσε να εφαρμόσει το, τις διατάξεις για το έγκλημα το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 416 του ποινικού κώδικα, το έγκλημα συμμετοχής σε, σε οργανώσεις ε, που έχουν χαρακτήρα μαφίας, καθορίζω, εντοπίζοντας τον τρόπο λειτουργίας αυτών των, οργανώσεων, που είναι καθαρά μαφιόζικος τρόπος, διότι μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με την πολιτική εξουσία και να ενταχθεί, να μπει, αν θέλετε, και στην ε, οικονομία της ε, πρωτεύουσάς μας. Η μαφία δεν έχει σύνορο, παρά μόνο τα, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να ε, καθορίσει την ζωή των πολιτών και την οικονομία των χωρών μας. Θέλουμε να ζητήσουμε σε όλη την Ευρώπη να μην ε, ε, πέσει στο στα σφάλματα, να μην επαναλάβει τα σφάλματα τα οποία κάναμε εμεί ορισμένε ε, περιοχέ που αρνήθηκαν τα εγκλήματα τη ε, μαφία, στο Μιλάνο, σε κάποιε περιοχέ ε, του Βορρά, διότι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα τη Σικελία, τη Καλαβρία και τη Καμπανία για να βρεθούν εκ των υστέρων μετά από κάποια χρόνια με πραγματικές ε, οργανώσεις που είχαν ε, εγκατασταθεί στις πόλεις τους ε, που μπορούσαν να επηρεάσουν τις δημοτικές και πολιτικές εκλογές και να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη. Η μαφία δεν έχει σύνορα και δεν θα πρέπει να έχει και σύνορα η καταπολέμηση της μαφίας. Θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε την μαφία. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι ένα κακό βαθιά ριζωμένο ε, στην ε, Ιταλική οικονομία, στην Ευρωπαϊκή οικονομία και στην οικονομία όλου του κόσμου. Από την άλλη πλευρά, αυτά ήταν τα συμπεράσματα της ε, ειδική Επιτροπής για, το οργανωμένο έγκλημα για τη διαφθορά και για το ξέπλυμα του χρήματος, που είχε δημιουργηθεί από αυτό το, το κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία και στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 ολοκλήρωσε το έργο της ε, και κάναμε ένα ψήφισμα το οποίο δέχτηκε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, τις, ε, για την μαφία σε όλη την Ευρώπη και εκεί σε αυτό το ψήφισμα υπάρχουν και στην έκθεση υπάρχουν ε, συστάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις δραστηριότητες, ε, δραστηριότητες οι οποίες ελπίζω θα ενσερνιστεί όλη η Ευρώπη. Υπάρχει μια δουλειά που έχει γίνει, την οποία σας την παραδίδουμε και που έχει σαν στόχο να ε, θέσει ενώπιον των ευθυνών της τη χώρα μου καταρχάς, διότι απέναντι σε κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει ήδη η Ευρώπη έχουμε καθυστερήσει, ασυγχώρητα καθυστερήσει. Στην ε, ε, ενσωμάτωση κάποιων οδηγιών στη χώρα μας και να τις εφαρμόσουμε. Ε, έχουμε επιταχύνει την, ε, δραστή οδηγία του, 2016, του 2006, συγγνώμη, διότι την, που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών κατάσχεσης και Επίσης ε, στον, ε, στον νόμο του 2014 ε, μπορούμε να μπορούμε, έχουμε ενσωματώσει μάλλον στην Ιταλική νομοθεσία τα θέματα της, που αφορούν την οδηγία που αφορά την αναγνώριση των κάποιων εγκλημάτων. Δηλαδή, σε κάποιου τομεί έχουμε κάνει το καθήκον μας, σε, κάποιες, σε κάποιους άλλους τομείς όχι. Και πιστεύω ότι η δουλειά αυτή την οποία κάναμε στην ε, Επιτροπή μας ε, και τώρα που ολοκληρώνεται η Ιταλική Προεδρία, μπορούμε να σας ζητήσουμε κάποιες, να αναλάβετε κάποιες ευθύνες ε, και να υιοθετήσετε κάποιες διατάξεις. Όπως είπε και ο πρόεδρος, τον οποίο ευχαριστώ, όταν μου έδωσε το λόγο, υπογράμμισε κάποιες, κάποια θέματα για τα οποία εργάζεται το Κοινοβούλιο αυτό και ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης που θα συνεδριάσει αυτές τις μέρες θα υιοθετήσει τις αντίστοιχες αποφάσεις όπως ελπίζουμε ότι και το τελευταίο Συμβούλιο της Ιταλικής ε, Προεδρίας θα δώσει έμφαση σε, αυτή την, σε αυτόν τον πόλεμο. Και στην, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει γρήγορα να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό προτείνουμε επίσης. Θέλουμε ε, το γραφείο του Ευρωπαίου εισαγγελέα να αποτελέσει μια υπηρεσία που θα οδηγεί τον πόλεμο κατά τις ε, μαφίες όλες οι έρευνες ε, για, τα, για τις έρευνες για όλες οι έρευνες που γίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη για τις δραστηριότητες που έχουν χαρακτήρα μαφίας να ε, κατευθύνονται από αυτή την ε, ε, εισαγγελία. Επίσης να υπάρχει μια διαδικασία κατάσχεσης που θα συμπληρώνει την αντίστοιχη οδηγία, οδηγία την οποία θεωρούμε ένα βήμα πρόοδου, λαμβάνοντας όμως την υπόψη την εμπειρία της χώρας μας, τα μεγάλα αποτελέσματα που είχαν τα προληπτικά μέτρα, θέλουμε η όλη διαδικασία της κατάσχεσης να γίνεται και απουσία ποινική καταδίκης, έτσι ώστε να, να αναγνωρίσει και την Ιταλική πρακτική που εφαρμόζουμε εμείς. Αυτοί που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους την, τον πόλεμο για τη μαφία, οι εισαγγελείς παραδείγματος χάρη της Σικελίας, του Παλέρμου, ο Μπορσελίνο, ο Φαλκόνε ε, μας έμαθαν, μας δίδαξαν ότι η μαφία κυνηγάει το χρήμα και κάνει τα πάντα για να κερδίσει το χρήμα. Και επομένως αυτό το οποίο φοβούνται περισσότερο είναι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα τους στερήσουν τα χρήματα αυτά τα οποία θα τους επιτρέψουν ε, να ε, ε, χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Πρόσφατα, σαν Επιτροπή, προσφέραμε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο μία πρόταση αναθεώρησης ριζικής της νομοθεσίας μας, διότι θεωρούμε ότι μετά από κάποια χρόνια πειραματισμού γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα αποτελέσματα ε, στα θέματα κατάσχεσης ε, ε, του προϊόντος της μαφίας και το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε τα αγαθά αυτά στην κοινωνία, διότι δεν είναι μόνο να τα πάρουμε από, τους, από, την, από τη μαφία, αλλά να τα επιστρέψουμε και στην κοινωνία διότι βίαια τα πήρανε τα αγαθά αυτά από έντιμους πολίτες και το κράτος πρέπει σε αυτούς να τα επιστρέψει, διότι προσφέρουν εργασία, ανάπτυξη και ε, επιτρέπουν να ξεπεράσουμε τις, ε, όλες αυτές τις διαφορές ε, και τις ανισότητες που δημιουργεί η μαφία στις χώρες μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ε, να προτείνει μια νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει συγκεκριμένα την έννοια ε, της εγκληματικής, ε, των εγκληματικών δραστηριοτήτων οργανώσεων που συνδέονται με την μαφία. Και αυτό που θα ισχύει για όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, να σας δώσω τα, τις έρευνες που γίνονται από την εισαγγελία της Ρώμης για να ε, καθορίσουμε μία δραστηριότητα μαφιόζικη δεν θα πρέπει απλώς και μόνο να συνδέεται με κάποιες μάρκες, με κάποια ονόματα τα οποία είναι γνωστά, αλλά θα πρέπει να ε, εντοπίσουμε τις διαδικασίες, τις μαφιόζικες διαδικασίες που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη οργάνωση. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως πριν από την ε, πρόταση για την οδηγία για, την, ε, για το ξέπλυμα του, του χρήματος, ε, μία, μία πρόταση γενικότερη όσον αφορά το ξέπλυμα και έτσι ώστε να ισχύει μία ενιαία νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα στη χώρα μας αυτό βέβαια δεν έχει φέρει αποτελέσματα και προχωράμε και ζητάμε με πάρα πολύ ε, ταπεινό τρόπο την, ε, την πρόταση αυτή. Η, η ικανότητα της μαφίας είναι ότι μπορεί να κινείται σε δύο τροχές. Το ένα είναι ότι κάνει οι παράνομες δραστηριότητες, κερδίζει χρήματα και από την άλλη πλευρά τα χρήματα αυτά τα επενδύει στην κανονική οικονομία. Και αυτό το ξέπλυμα του χρήματος είναι δηλαδή ε, είναι η συνοσυνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις δύο τροχές. Επίσης, ε, πρέπει να κάνουμε προτάσεις και να ισχύσει μια νομοθεσία όσον αφορά την παρακολούθηση των ε, τηλεφωνικών κλήσεων. Γιατί και αυτό είναι ένα στοιχείο, ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να πολεμήσουμε την μαφία. Επίσης ζητάμε να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναρμονισμένα ή συντονισμένα μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουμε την διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και αναφερόμαστε παραδείγματο χάρη ε, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, των εξαποστάσεως κυρίως, κυρίως όσον αφορά το βίντεο πόκερ και, τις, και, τα, συστή, και τα στοιχήματα. Και θέλουμε να υιοθετηθούν κοινέ γραμμές για να αναγνωρίζουμε τον επαγγελματισμό και την εντιμότητα όλων όσων εμπλέκονται σε αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Επίσης θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει πιο ομογενές το σύστημα ε, ορισμού των διαφόρων ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών οργανώσεων. Ε, ήδη έχει υιοθετηθεί μια κάποια νομοθεσία στο παρελθόν, αλλά ακόμα δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόσει την νομοθεσία. Γιατί και με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει σωστά η έρευνα και η η εξακρίβωση ε, της νομιμότητας όλων αυτών των οργανώσεων και της κατάσχεσης ε, κάποιων αγαθών κατάσχεσης προϊόντος εγκλήματος. Θέλουμε επίσης ε, να προωθήσουμε την πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι αστυνομικέ δυνάμεις της Ιταλίας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κατά της μαφίας. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Και σε αυτή την επιτροπή, την οποία θέλουμε να καταθέσουμε την εργασία μας, και θέλουμε να καταθέσουμε και τα αιτήματά μας έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την θητεία να αποκτήσει μια ειδική επιτροπή η οποία να είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της ε, εγκληματικής δραστηριότητας ε, ε, που έχει χαρακτήρα μαφίας. Ε, να έχει ένα εργαλείο τέλος πάντων, να αποκτήσει ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει να, έχει, να δώσουμε τη συγκεκριμένη και ε, την αρμόζουσα ε, προσοχή στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, ίσως καταχράστηκα λίγο και του χρόνου σας, αλλά τέλος πάντων ήταν ίσως και απαραίτητο να σας δείξω με λεπτομέρειες και την εργασία μας, αλλά και τις απόψεις μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Ρόζη. Και δεν καταχράστηκε του χρόνου μας, γιατί έχουμε αφιερώσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της σημερινή διάταξη της συζήτησης του θέματος αυτού. ήθελα ίσως ε, να μας δώσει πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά θεώρησα καλύτερο τελικά να ακούσουμε και τις απόψεις των συναδέλφων για να έχουμε μετά και μια συζήτηση. Στην αρχή είπε ότι από, το, από πότε ήσουν εδώ από το 89 στο 94 ευρωβουλευτής, πριν τη Λισαβόνα δηλαδή. Και είδατε μετά τη Λισαβόνα πόσο πολύ νομοθεσία έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε στον τομέα αυτό. Είναι εξαιρετικό αυτό το επίτευγμα. Μπορεί να έχουμε πολιτικές ε, διαφορές μεταξύ των συναδέλφων. Πάντως συμφωνία ε, γενική υπάρχει. Εξού και η Επιτροπή ΚΡΙΜ ε, που ανέφερες ε, και παρά τη διαφωνία μας, επαναλαμβάνω, καταφέρνουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Έχουμε και τον Κλάντιο, Κλάντιο Φάβα εδώ που ήταν μέλος της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Ανέφερες και εσύ βέβαια και άλλους συμμετέχοντες. Ήταν τεράστιο το έργο της Επιτροπής Αυτά που κάνετε εσείς βέβαια είναι σημαντικά, δεν είναι μόνο ένα πρακτικό νομοθετικό καθήκον, επηρεάζει και την ίδια την κοινωνία. Η Εξεταστική σας Επιτροπή βέβαια διαδραματίζει ε, κοινωνικό, μάλλον παράγει κοινωνικό έργο όπως είπα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχει απλά το νομοθετικό καθήκον. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι εδώ πολύ πεπειραμένοι συνάδελφοι θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ορισμένοι ήταν και μέλη της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Ο Τίμωθη Κέρκοπ από την ομάδα ECR, συντονιστής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών, είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι είναι μια έκθεση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωταρχικά μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφαιρούν ένα κράτος μέλος, όμως είναι τεράστια η σημασία του πώς και τα υπόλοιπα κράτη αντιμετωπίζουν και τις νυν και τις μελλοντικές απειλές από εγκληματίες και τρομοκράτες. Ήμουν μέλος της Επιτροπής ΚΡΙΜ, ε, έχω σπουδάσει νομική, το ξέρετε φαντάζομαι, και υπάρχουν ζητήματα εδώ θα ήθελα να τα υπογραμμίσω γιατί φαίνεται ότι θα μπορούσαν να, εφαρμόζονται για όλους μας, για ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, θα ξεκινήσω με τα επίπεδα συνεργασίας, όπως αναφέρεται και στα πορίσματα της έκθεσης και της ε, μικτής ερευνητικής ομάδας. Με ενδιαφέρει αυτό το θέμα των μικτών ερευνητικών ομάδων γιατί με τη δική μου έκθεση συγκροτήθηκαν αρχικά αυτές οι ομάδες. Και έκτοτε, όταν πέρασε δηλαδή η έκθεση και μετά, ε, μου δημιουργήθηκαν κάποιες ανησυχίες ε, γιατί ναι μεν καλές οι προθέσεις, ε, αλλά πρακτικά δεν έχουμε σημειώσει επαρκή πρόοδο, δεν έχουμε επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών ε, με τις ε, διάφορες ε, αρχές επιβολής της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Μπορεί να κάνει ό,τι κάνει για τη μαφία η Ιταλία, που δεν είναι όμως κάτι που αφορά μόνο την Ιταλία. Θα μπορούσαν να το υιοθετήσουν για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος σε άλλες χώρες και γι' αυτό θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Έρχομαι τώρα σε ένα σημείο το οποίο, εκτός αν δεν το διάβασα πολύ προσεκτικά, δεν φαίνεται να ε, αποδίδει έκθεση τόσο μεγάλη σημασία όσο θα ήθελα εγώ τουλάχιστον. Μιλώ για ε, το κυβερνό έγκλημα. Έχουμε τις νέες τεχνολογίες, νέους τρόπους με τους οποίους οι εγκληματίες μπορούν να, να ασκούν τις δραστηριότητές τους. Ε, για μένα όμως, σχεδόν η μεγαλύτερη απειλή σήμερα είναι η χρήση του διαδικτύου και το κυβερνό έγκλημα. Έχουμε δει πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα προσφάτως, όχι μόνο από εγκληματικές δραστηριότητες ε, της μαφίας ή άλλων εγκληματικών οργανώσεων, Έχουμε δει όμως και μεταξύ κρατών ή σε κράτη. Για παράδειγμα, πώς εξελίσσεται η παγκόσμια πολιτική στις μέρες μας. Νομίζω ότι ε, και οι κυβερνοαπειλές χρησιμοποιούνται δυστυχώς εναντίον των εμπορικών, πολιτικών συμφερόντων και των δικών μας ε, οργάνων. Είχαμε κάποιες πρωτοβουλίες στο Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε μίζων εγκλήματα και διαπιστώσαμε όμως ότι οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες προηγούνται είναι ένα βήμα πιο μπροστά από μας σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές ε, μεθόδους που χρησιμοποιούν. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή κρίμη και θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Η ε, επανασύσταση αυτής της Επιτροπής είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Οποιαδήποτε όμως πίεση επιρροή από τους συντάκτες ε, της θα βοηθούσε πάρα πολύ ω προ αυτό. Τέλο, ό,τι αφορά το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Οι αρχέ επιβολή ομοθεσία και εμεί διαφωνούμε εδώ και ε, καιρό σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση αναγνώριση πριν την κατάσχεση, την δίμευση. Υπάρχουν λοιπόν περσιακά στοιχεία που σχετίζονται ε, και με την καθαρή θέση ή και με ε, δηματικές δραστηριότητες. Πώς θα διαχωρίζουμε αυτά τα δύο αυτό πρέπει να το δούμε και μετά να προχωρήσουμε στην κατάσχεση. Ευχαριστώ. Έχουμε 8 συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο από την Επιτροπή. Αν δεν τηρήσουμε το δίλεπτο, δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους ε, Ιταλούς συναδέλφους για να σχολιάσουν. και θα προλάβουν αν περιοριστούμε στο δίλεπτο. Κατερίνα Τζίντσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να κρύψω τη συγκίνησή μου που μου επιτρέπεται να μιλήσω ε, σε αυτή την ε, συνεδρίαση. Και η κυρία Μπίντι και ο πρόεδρος ε, αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά. Ε, εμένα όμως αυτά τα θέματα με έχουν θίξει και οικογενειακά. Ε, γι' αυτό είμαι και τόσο συγκινημένη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οργανωμένη εγκληματικότητα ε, ξεκίνησε μπορεί από την Σικελία, αλλά με τα χρόνια έχει, έχει τροποποιηθεί, έχει αλλάξει και έχει εγκατασταθεί σε όλη την χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε, να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέτρο για να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ την πρόεδρο Μπίντι που θέλησε να παρουσιάσει αλλά αυτόν τον τόσο ολοκληρωμένο τρόπο την ε, εργασία της Επιτροπής ε, της Γερουσίας και της Βουλής για τις δραστηριότητες της μαφίας και, άλλων, ε, και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Μία μέθοδο που, που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι, η κατά της μαφίας είναι να την αποδυναμώσουμε οικονομικά ε, εφαρμόζοντας ε, αποτελεσματικά τα μέτρα της ε, κατάσχεσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες και τα προϊόντα των εγκληματικών δραστηριοτήτων επηρεάζουν άμεσα την οικονομία των χωρών μας. Η Ιταλία έχει συγκεκριμένη εμπειρία για τα θέματα αυτά, η Σικελία πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν έρευνες του Πούλα Αντιμάφιε ε, που ξεκίνησα από τον πατέρα μου, ο οποίος σκοτώθηκε το 1983 στις ε, πρώτες, ε, ε, στις, στις πρώτες προσπάθειες που κάναμε και τον ακολούθησαν 9 χρόνια μετά ο Μπορσαλίνο και ο Φαλκόνε που σκοτώθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους. Λοιπόν, ξεκίνησε ανα τα θέματα, ε, ξεκίνησε μάλλον και η δημιουργία και οι προσπάθειες ε, αντιμετώπισης ε, των δραστηριοτήτων της μαφίας σε οικονομικό επίπεδο και από έναν άλλον εισαγγελέα ο οποίος σκοτώθηκε μερικούς μήνες, ένα χρόνο πριν από τον πατέρα μου. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά πράγματα και στην Ιταλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο με το Τάμπερε, τα συμπεράσματα του Τάμπερε το 2009 και καταλήξαμε στην οδηγία της 3ης Απριλίου του 2014 όσον αφορά το πάγωμα και τις κατάσχεσης ε, προϊόντων εγκλήματος. Η οδηγία θα αντικαταστήσει την απόφαση πλαίσιο του Φεβρουαρίου του 2005 εισάγοντας κάποιες διατάξεις που από τη στιγμή που θα εφαρμοθούν θα επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε ε, αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Λυπάμαι, αλλά δεν ήμουν και τότε βουλευτής ε, τώρα έγινα βουλευτής, που δεν συμμετείχα στις ε, δραστηριότητες της Επιτροπής ε, Κρίμα, που πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην, όλη προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Ευχαριστώ τον κύριο Κίρκοφ για τη δουλειά που έχει κάνει και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ολοκληρώνω συμμερίζοντας όλα τα συμπεράσματα τα οποία παρουσίασε η κυρία Μπίντι για τις ε, δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα ήθελα για άλλη μια φορά να ε, σταματήσω στο οικονομικό θέμα, γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ασκήσουμε στον το μεγαλύτερη πίεση και στα εθνικά, ε, σε εθνικές θεσμικά όργανα, έτσι ώστε να υιοθετηθούν όλα τα απαραίτητα κείμενα εγκαίρωσο και θα πρέπει επίσης να εγκριθεί να εγκριθούν ε, και κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ζητάμε από, το, από την Επιτροπή να ε, προτείνει ε, κάποια μέτρα και να υιοθετήσει μέτρα, παραδείγματος χάρη, όπως η κατάσχεση πριν από την ποινική καταδίκη. Αυτός είναι ένας δρόμος τον οποίο όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε, προωθώντας ε, την ε, νομοθεσία που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο την εγκληματική, τις εγκληματικές δραστηριότητες σε κάθε μορφή που έχουν αυτές ε, και σε κάθε πλαίσιο που υιοθετούν και είναι ένα καθήκον που έχουμε όλοι μας διότι πραγματικά έχουν θυσιαστεί πολλές ανθρώπινες ζωές στην προσπάθεια αυτή. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Κατρίνα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Ο κύριος Τόμας Σιτόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω Ιταλικά, αλλά δεν μιλάω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θα μιλήσω τσέχικα. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση. Πρόσφατα, πολλή συζήτηση έχει γίνει για τη συμμετοχή της Ιταλικής Ισικελικής μαφίας στο λαθρεμπόριο ανθρώπων ε, στην Ιταλία. με επιδότηση μάλιστα. Και ε, αναφέρεται ότι η Ιταλική μαφία κάνει εκτροπή επιδοτήσεων που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους ε, πρόσφυγες στο νότο της Ιταλίας. Έχετε κι εσείς παρόμοια πληροφορία και τι θα κάνετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί διαφάνεια ε, σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων. Αυτό βοηθάει ενδεχομένως. Ευχαριστώ Τόμας και για την συντομία σου. Επόμενος ο ε, Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Κρίμ όταν αυτή είχε συσταθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μπίντι. Εδώ είμαι δεν βλεπόμαθα για πρώτη φορά. Βρεθήκαμε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξανά. Ευχαριστούμε πολύ που μας μεταφέρατε την Ιταλική εμπειρία του Ιταλικού Κοινοβουλίου εδώ. Μία ερώτηση σύντομη. Καταρχάς, ποιο θα ήταν το πιο σαφές μήνυμα, μάθημα θα έλεγα, όσον αφορά τον εισαγγελέα, τον, Ευρωπαϊ... τον Ευρωπαίο εισαγγελέα. Η επιλογή της, ε, η, δημιουργία, η... θέλουμε να δούμε ποια θα συγκρίνοντας ε, ε, τα όσα έχουν γίνει στην Ιταλία όσον αφορά τις δραστηριότητες ε, της Ιταλικής εισαγγελίας κατά της μαφίας, πώς θα μπορούσαμε να διδαχτεί, θα μπορούσαμε να διδαχτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για, τον Ευρωπαίο εισαγγελέα κατά της μαφίας και όσον αφορά την μορφή αλλά όσον αφορά και τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες που θα έχει. Δεύτερον, να επαναλάβω αυτό που είπε, που είπε και ο συνάδελφος Τίμωθη Κίρκοπ για τις ε, ερευνητικές ε, ομάδες, τις Joint Investigation Teams. Τι, ποια είναι η αξιολόγηση σας ε, όσον αφορά την λειτουργικότητα αυτών των ομάδων. Πώς δηλαδή λειτουργούν στην διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση των, του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα να είσαστε ειλικρινείς στο σημείο αυτό. Πώς αξιολογήθηκε από την Επιτροπή η Ιταλική δέσμευση, η συγκεκριμένα η Ιταλική δέσμευση σε αυτές τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες και ποια είναι τα διδάγματα όσον αφορά την νομοθετική, το νομοθετικό έργο και τις νομοθετικές προτάσεις που θα μπορούσε να υποβάλει αυτή η Επιτροπή μας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ε, δημοσίων ελευθεριών. Διότι ασχολούμεθα με την ποινική νομοθεσία, με τις, ε, με τις δικονομίες, με τις ποινικέ, με την ποινική δικονομία και θέλουμε να ξέρουμε εμείς σαν νομοθέτες στο ποινικό επίπεδο τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση. Αλεξάνδρα Βασιλή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόεδρο Μπίνδη για την, και τη συγχαίρω για την ακρίβεια αυτής της έκθεση. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια σωστή ε, πλατφόρμα για τις εργασίες της Επιτροπής, λαμβάνοντας ε, υπόψη τις προτάσεις που γίνονται. Θα ήθελα να ε, σταματήσω σε κάτι το οποίο είναι κοινό ίσως, αλλά είναι σημαντικό. Όταν ε, υιοθετούμε ε, ή όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές οδηγίες, θα πρέπει να ε, απλουστευτεί η διαδικασία ε, μεταφοράς των οδηγιών αυτών σε εθνικό δίκαιο. Επίσης πρέπει να είναι και απλουστευμένη η γλώσσα ε, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εφαρμογή και η ερμηνεία που δίνεται σε εθνικό επίπεδο να είναι εις βάρος της οδηγίας. για το, το, το, πρόσφατο, τα πρόσφατα κείμενα τα οποία υιοθετήθηκαν ε, για τις ε, εγκληματικές δραστηριότητες ε, που έχουν χαρακτήρα μαφίας, εκεί ο ορισμός δεν ήταν σαφής και αυτό ήταν εις βάρος του κειμένου. Επομένως θα πρέπει και η Κομισιόν να, έχει, να προτείνει συγκεκριμένους και σαφείς ορισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μαφία δεν είναι ιταλικό προϊόν μόνο δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ιταλίας. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας και να λέμε αυτό, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα, για ένα δράμα ε, ευρύτερο, το οποίο καταστρέφει οι ε, οικογένειες ολόκληρες με τα τυχερά παιχνίδια κτλ. Υπάρχουν στην Ιταλία στο εξωτερικό, και στο εξωτερικό. Επίσης αναφέρθηκε ε, το θέμα της, ε, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενιαίος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Αυτό είναι πήγον. Ο συνάδελφος μίλησε για μια κοινή ερευνητική ομάδα, η υπέρ, που και αυτό ε, συνάδει με την αρμοδιότητα, αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και κυρίως όσον αφορά, πρέπει να προχωρήσουμε και όσον αφορά και την κατάσχεση αλλά και την, ε, την απόδοση των προϊόντων αυτών, των κατασχεμένων προϊόντων. Η Μπίργκη, η συντονίστρια της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την έκθεση από τη συνάδελφο Μπίντι που έδειξε σαφέστατα ότι το οργανωμένο έγκλημα πράγματι είναι κάτι που υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Παράλληλα νομίζω ότι ξεκαθαρίζει η έκθεση αυτή ότι υπάρχουν και εθνικές διαφορές στο οργανωμένο έγκλημα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που γίνονται, η σύνδεση οργανωμένου εγκλήματος ε, και ε, του νομικού χώρου ε, οι διαφορές στις δημόσιες διοικήσεις, οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Γι' αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε τη χρυσή μέση λύση, τη χρυσή οδό για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν και κοινά σημεία που τα αναφέρατε και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για την καταπολέμηση της απάτης και του ξεπλήματος χρήματος. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία. Τώρα, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Το πιο σημαντικό για αυτή την Επιτροπή είναι να παρακολουθεί όλες τις οδηγίες και τα μέτρα που έχουμε ήδη θεσπίσει και αυτά που αποφασίσαμε και θεσπίσαμε κατά την προηγούμενη θητεία γιατί θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά και να καταστούν αποτελεσματικά πριν αρχίσουμε με νέες διαδικασίες και μέτρα. Τέλος, νομίζω ότι όλα τα μέτρα που αποφασίζουμε εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι αποτελεσματικά μόνο αν τα κράτη-μέλη μας είναι πρόθυμα να τα εφαρμόσουν και να συνεργαστούν. Ίσως ε, η συνάδελφος Μπίντι μπορεί να το σχολιάσει αυτό γιατί ανησυχούμε ότι τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα κράτη-μέλη και δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε πολύ αποτελεσματικά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, ούτω ώστε το πλαστάσιό μας να γίνει αποτελεσματικό πριν προβούμε στη λήψη νέων μέτρων. Αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος συνέχισης του έργου μας. Ευχαριστώ δηλαδή μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μπίντι και ευχαριστώ και για την παρουσία σας αλλά και για την ε, παρουσίαση που μας κάνατε. Χάρηκα ιδιαίτερα που σας άκουσα να μιλάτε για την ανάγκη να αναγνωριστεί και η μαφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί ακόμα και σήμερα πολλά κράτη-μέλη αρνούνται την παρουσία μιας οργανωμένης εγκληματικότητας μαφιόζικου χαρακτήρα και σε άλλες, άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή θεωρούν ότι ένα, πρόκειται για ιταλικό προνόμιο, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Χάρηκα επίσης που σας άκουσα να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά της μαφίας. Χάρηκα διότι όταν τον Ιούλιο ε, ε, υποδεχθήκαμε τον κύριο Ορλάντο, τον Υπουργό Ορλάντο και όταν τον ρώτησα εάν χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ε, ευρωπαϊκή εισαγγελία κατά της μαφίας όπως το δικό μας το ιταλικό μοντέλο της ΔΙΑ μου είπε ότι είναι ένα μοντέλο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ότι, ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Λυπήθηκα τότε, χαίρομαι τώρα όμως που, λέ, που τώρα έχουν αλλάξει ε, τα πράγματα, διότι η, δημιουργία μιας ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, θα οδηγήσει και σε μια ε, ομοιογένεια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δηλαδή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί κάπως η, η Ευρωπαϊκή Νομολογία έτσι ώστε να επιτρέπεται και η δίωξη αλλά και η συνέχιση των ερευνών και διαρωτώ με μήπως ε, ανάμεσα στις άλλες προτάσεις ε, που υποβάλλεται όσον αφορά την κατάσχεση, το ξέπλυμα ε, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μήπως θα μπορούσαμε να συμπεριλαμβούμε και την, την πρόβλεψη της καθυστερημένης κατάσχεσης ή καθυστερημένης σύλληψης όσον αφορά την, την αναδρομική ίσως, ναι, όπως ισχύει και στην Ιταλία για να μπορέσουμε να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να προχωρήσουμε στην έρευνα, να βρούμε τις, τους πραγματικούς εγκληματίες και να μην σταματήσουμε στο μικρό ψάρι ας πούμε. Δηλαδή να μην, να μην συλλάβουμε ε, αυτόν ο οποίος διαπράττει τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο αδίκημα, αλλά να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε αυτούς που τον καλύπτουν και που τον στηρίζουν. Είπατε ότι η όλη καταπολέμηση, τα, με τα θέματα της ε, κατάσχεσης ε, και της απόδοσης του προϊόντος του εγκλήματος στο, την κοινωνία, στους πολίτες, καθυστερεί. Υπάρχουν πάρα πολλά χιλιάδες κτίρια στην Ιταλία τα οποία έχουν κατασχεθεί, αλλά η όλη η διαδικασία επιστροφής των αγαθών αυτών στους νόμιμους ιδιοκτήτες καθυστερεί. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια Υπάρχει και το, η ψυχολογία ε, των πολιτών που παραδείγματο χάρη ε, στην Ιταλία δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα κτίριο το οποίο ανήκει σε ένα μαφιόζο. Αλλά τέλος πάντων για να ολοκληρωθεί ε, το όλο έργο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, δηλαδή για την επιστροφή των ε, αγαθών αυτών, ίσως θα έπρεπε να το συμπληρώσουμε και να πούμε ότι τα, ε, τα αγαθά αυτά θα πρέπει να αποδοθούν σε κάποια ιδρύματα, ευαγή ιδρύματα κτλ όπως επίσης για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, οι μαφιόζικες δραστηριότητες επηρεάζουν και την διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Και συμφωνώ με την κυρία Μουσολίνη ότι θα πρέπει να ε, δημιουργηθεί ξανά, να συσταθεί ξανά η Επιτροπή Κρίμα. Πραγματικά δεν θα πρέπει όλα αυτά τα μέτρα που εδώ συζητάμε να παραμείνουν νεκρό γράμμα. Ευχαριστώ. Έχω δώσει αρκετό χρόνο στους συναδέλφους γιατί γνωρίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω όμως να δώσω και στους Ιταλούς ε, ε, συναδέλφους κάποιο χρόνο από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Πρώτα λοιπόν να ολοκληρώσουμε με τους δικούς μας συναδέλφους. Η Εύα Ζολή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την πρόεδρο της ε, Ιταλικής αυτής ε, Εκταστικής Επιτροπής που ήρθε εδώ για να μοιραστεί την εμπειρία της. Έχω ε, την ανάγκη να πω κάτι πολύ απλό. Δεν ακούμε κάτι καινούριο ή κάτι άγνωστο. Η Ιταλία έχει πολύ ικανούς εισαγγελεί και δικαστικού, που δεν είναι όμως αρκετοί τον ρυθμό γιατί δεν υπάρχει ε, στον προπολογισμό η απαιτούμενη προτεραιότητα για τη δικαιοσύνη. Είναι λιγότερη... Ε, ε, έχετε τρεις εισαγγελείς Ε, το μισό από τη Γερμανία, το 1 πέμπτο από την Νορβηγία, 71 ευρώ κατά κεφαλήνα είναι για τη δικαιοσύνη στον προπολογισμό και είναι πραγματικά άθλημιστή των εισαγγελέων και των δικαστικών. Έχετε λοιπόν ε, τους ε, πολύ ε, καλούς αυτούς επαγγελματίες, δεν τους δίνετε όμως μέσα στην διάθεσή τους και δεν λύνονται τα προβλήματα με κείμενα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι έχετε κάνει για να τεθεί ένα τέρμα στην φιόζικη περιβαλλοντική κλιματικότητα που βάζει σε κίνδυνο την υγεία του πληθυσμού. Μιλώ για την Νότια Ιταλία ε, και για τα βουνά επικίνδυνων αποβλήτων ε, και απορριμμάτων τα οποία εκεί διατίθενται χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο εισαγγελίε τη Νάπολη. Πότε θα ξεκινήσουν δραστηριότητε, διαδικασίες για να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Ίσως ένα μέσο για να μπορέσετε εσεί να αυξήσετε τον προϋπολογισμό στη δικαιοσύνη. Θα ήταν να δείτε ε, τα στοιχεία από το LuxLeaks που δείχνουν ιταλικές εταιρείε που δεν πληρώνουν φόρους γιατί έχουν την στο Λουξεμβούργο. Δισεκατομμύρια θα μπορούσατε αυτά να τα δώσετε για τη ε, δικαιοσύνη, για το τομέα της δικαιοσύνης. Θα έπρεπε ίσως να δώσει η κυβέρνησή σας οδηγίες στις εφορίες για να δουν τι γίνεται με αυτές τις εταιρείε. Αλλιώς ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ γιατί ξέρουμε ότι το ποινικό δίκαιο δεν είναι καλά προσαρμοσμένο ε, για την δίμευση των περισσότερων στοιχείων των μαφιόζων και γι' αυτό έχετε βάλει και το θέμα της αστικής, έχετε δεχτεί την αστική δίμευση. Στη Γαλλία έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Χρειάζονται εθνικές μεταρρυθμίσεις για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά βασίζω πολλά ε, στην ε, στήριξη της Ιταλικής Προεδρίας και της Ιταλίας εν γέννη για την πρόθεση της οδηγίας για την απάτη, που είναι η βάση για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Και μέσω του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και της οδηγίας αυτής, ένα μέρος του αγώνα κατά της μαφίας θα έχει ξεκινήσει. Γιατί μιλάμε και για προσβολή των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Μπίντη, θα σας δώσω τώρα το λόγο Θα ήθελα να σας ε, ε, παρακαλέσω να δώσετε και το λόγο στους συναδέλφους σας όμως, να μου πείτε εσείς ε, σε ποιους λοιπά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Θα συζητήσω εν συντομία μαζί τους γιατί θα ήθελα και οι άλλοι ε, τα άλλα μέλη της Επιτροπής, η κυρία Γκαραβίνη παραδείγματος χάρη, η οποία προεδρεύει της Επιτροπής ε, ε, για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων της μαφίας σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, που ήταν και η συγγήτρια της έκθεσης που τη ζητήσαμε, θα μπορέσει να σας δώσει και κάποιες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ετέθησαν. Και θα ήθελα να ζητήσω και από τον Αντιπρόεδρο Φάβα να πάρει το λόγο. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν και αντιπρόσωποι των άλλων ε, πολιτικών δυνάμεων, όλων των πολιτικών δυνάμεων που, ε, που συμπεριλαμβάνονται στην Επιτροπή. Η κυρία Σκοπελίτη και εκεί ο μπαμπάς, ο πατέρας ήταν δικαστικός και, που, και πλήρωσε με τη ζωή του τον πόλεμο κατά της Ντράγκετα. Κύριος Πολέτη επίσης. Ε, υπάρχουν, έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες ε, και σε αστυνομικό και σε δικαστικό επίπεδο που μας οδήγησαν σε κάποιες επιτυχίες. Ε, Διλέλο, σοσιαλιστής γραμματέας της Επιτροπής και ο κύριος Ντούβα που είναι ο επικεφαλής ε, της ομάδας ε, των πέντε αστεριών στην Επιτροπή και ο κύριος Ζαρούσο. Και αυτός από τα 5 Stella, τα πέντε αστέρια. Και αν θέλουν να πάρουν το λόγο Γκαραβίνη, Φάβα ή τέλος πάντων μπορούν να συμπληρώσουν την ε, παρέμβαση που θα είναι σύντομη. Το ένα είναι ότι συμμερίζομαι απόλυτα Λίγα λεπτά, λίγα λεπτά εγώ θα απαντήσω και μετά θα είναι οι συνάδελφοι. Να πω ότι συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε η κυρία Σίμπελς, ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τις οδηγίες, τα στις διατάξεις ε, που θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε. Όλες ε, οι χώρες έχουν καθυστερήσει και η χώρα μου επίσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε με θάρρος και να... Αυτά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει θεωρητικά να τα κάνουμε και πρακτικά. στο θέμα της δικαιοσύνης εν γέννη στη χώρα μου να πω ότι είναι αλήθεια ότι αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα λόγω της δημιουργίας αυτών των πουλ που, των, ομάδων, των κοινών ομάδων που ε, χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη κατά της ε, μαφίας. Ξεκίνησαν από τον Κινίτσι, τον Φαλκόνε, τον Πορσαλίνο και συνεχίζουν ακόμα. Δημιουργήσαμε, δημιουργήθηκαν ε, θέσεις εισαγγελέων, δικαστών, αστυνομικών που είναι αφιερωμένοι αποκλειστικά σε αυτό τον πόλεμο. Και δημιουργήθηκε και αυτή η Εθνική Εισαγγελία. Και από αυτή την οργάνωση έτσι όπως την έχουμε οργανώσει τώρα το, όλο σύστημα, μπορούν να αντιληφθούν και διδάγματα, όπως είπε ο κ. Αγγιλάρ, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πιστεύω ότι και ακόμα και στα, αποτελέσματα της μάχης κατά την μαφία πληρώνουμε τις καθυστερήσεις του δικαστικού συστήματος και πληρώνουμε την ε, έλλειψη μιας ε, ε, νομοθεσίας που δεν είναι τόσο απόλυτη και κατηγορηματική απέναντι σε κάποια αδικήματα, σε κάποια εγκλήματα. Εμείς ζητάμε να έχουμε στη διάθεσή μας πιο αυστηρά μέτρα για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει η μαφία, κυρίως η διαφθορά και όλα τα οικονομικά εγκλήματα και η, ε, ούτως ή άλλως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τυποποιήσει κάποια περιβαλλοντικά εγκλήματα και θα, είναι και θα έχουμε και την Ειδική Επιτροπή για τα απορρίμματα, για, για τα απορρίμματα. Ε, ούτως ή άλλως ε, πολλές χώρες έστειλαν τα, απόβλητά τους στη χώρα μας και στο, και στο παρελθόν με τις δραστηριότητες της Δράγκεντα και της Καμόρα. Και με τα ίδια μας τα τα χέρια δηλαδή καταστρέφουμε αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα τα οποία ε, παράγει η Ιταλική γη και ε, Έχουμε ξεκινήσει και τις δραστηριότητες ε, της Επιτροπής Έρευνες, μιας Επιτροπής για την ε, παράνομη ε, διακίνηση ανθρώπων. Δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομέρειες διαδικαστικές, αλλά ξέρουμε ότι η μαφία μπορεί να πάρει χρήματα και πόρους οπουδήποτε κι αν βρίσκονται αυτοί. Και σε μια πρόσφατη έρευνα στη Ρώμη ε, είδαμε ότι ε, εμπλέκονταν κάποιες ε, οργανώσεις που τοποθετούσαν τους μετανάστες σε κάποια στρατόπεδα και σε κάποια άλλα. Σίγουρα παρεμβαίνουν στις μεταφορές, ούτως ή άλλως δεν, υπάρχουν δημόσιο, δεν υπάρχει δημόσιο χρήμα το οποίο να μην μπορεί να πάρει η μαφία και να μην επωφεληθεί από οποιαδήποτε δυνατότητα που τη δίδεται. Και για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να πω τελικά ότι στα θέματα της κατάσχεσης, που είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα, έχουμε διμερείς συμφωνίες με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και θα θέλαμε αυτό να διευρυνθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες διότι Ξέρουμε ότι γίνονται και εμπλέκεται εδώ και οι, εμπλέκονται και άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία παραδείγματο χάρη. Και θέλουμε, θέλουμε να μπορούμε να, ας πούμε, κάποια ε, προϊόντα τα οποία, της, της δραστηριότητας της μαφίας που καταλήγουν εκεί, να μπορούμε να τα ε, πάρουμε πίσω. Να σας πω ότι όλα αυτά τα χωλάθη εντοπίσαμε κάποιες, κάποια ευαίσθητα σημεία ε, τα οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια Αλλά τέλο πάντων θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ε, συνεργαστούμε και με τι άλλε χώρε. Κυρία Καραβίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ουσιαστικά και όχι τυπικά την ε, πρόεδρο τη Επιτροπής κατά τη μαφία. διότι ε, επέλεξε να συζητήσουμε ε, και να εξετάσουμε τα θέματα των δραστηριοτήτων ε, της μαφίας σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι μια επιλογή πάρα πολύ σωστή Θα πρέπει να υπογραμμίσω κυρίως την αξία όλων αυτών, διότι είναι σημαντικό, ε, σημαντική και η παρουσία μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι δεν μπορούμε να ε, εξετάσουμε τα θέματα της ε, μαφίας <laughs> αυτή τη στιγμή, χωρίς να θεωρήσουμε ότι η μαφία είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Διότι τα φαινόμενα της μαφίας, που δεν είναι καθαρά ιταλικά, δεν είναι μόνο ιταλικά. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, διότι δείχνουν τη στενή συνεργασία ε, όλων αυτών των ε, εγκληματικών ε, οργανώσεων που είναι διαφορετικής προέλευσης αλλά που συνεργάζονται μεταξύ τους και η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία αντιμετώπιση συντονισμένη και σε ένα πνεύμα συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν, κυρίως για τον ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε συνεργασία με τις ε, εθνικές υπηρεσίες, αγγελικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την μαφία. Θα πρέπει να υπογραμμίσω επίσης ότι δημιουργήθηκε και στο ιστορικό της Επιτροπής μας η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάνω στην οποία εργαζόμαστε και η οποία γίνεται ευτυχώς ένας στόχος επιτεύξιμος και η Ιταλική Προεδρία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και έδωσε προτεραιότητα στα θέματα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, μία από τις επιθυμίες και τις ευχές της Επιτροπής μας είναι ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην περιορίζεται μόνο <coughs> σε μία έρευνα των διοικητικών ε, απατών αν θέλετε αλλά να γίνεται μια, ουσιαστικά μια εισαγγελία κατά την μαφία δηλαδή όχι μόνο να βλέπει διοικητικέ απάτες που σωστά είναι κακές και πρέπει να καταπολεμούνται α, όμως πρέπει να ε, ε, προσπαθεί να πετύχει συγκεκριμένους στόχους κατά της μαφίας. Να γίνει δηλαδή ουσιαστικά μια εισαγγελία κατά της μαφίας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά. Διότι με τον τρόπο αυτό, με την, όπως είχε πει και ο Τζοβάνι, Φαλκόνε τότε, θα δημιουργηθεί μία εισαγγελία η οποία θα συνδυάσει στοιχεία ε, που προέρχονται από διάφορες έρευνες, από διάφορες χώρες και έρευνες οι οποίες όμως στα, στις υποθέσεις, ε, τις εγκληματικές υποθέσεις και, στην, και στα κυκλώματα βλέπουμε ότι έχουμε ε, έχουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ε, από μια κοινή αρχή. Από μια κοινή αρχή. Άρα αυτά τα συμφέροντα, τα εγκληματικά και τα κυκλώματα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια ενιαία εισαγγελία. Με τη βοήθεια βέβαια των εθνικών εισαγγελιών κατά της μαφίας. Πιστεύουμε επομένως ότι αυτός πρέπει να είναι ένας από τους στόχους μας, στόχους ε, που πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πολεμήσουμε όσο, όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά την εγκληματικότητα. <clears throat> Και αναφέρομαι και στον κυβερνοχώρο ε, στην εγκληματικότητα ε, στον κυβερνοχώρο. Είναι μια δραστηριότητα πιο ευρεία ε, από πλευράς των εγκληματικών οργανώσεων Άρα και εκεί πρέπει να υπάρξει μια στενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, κυρίως συνεργασία ανάμεσα στις ερευνητικές αρχές. Αυτό το θέλουμε. Θέλουμε οι ερευνητικές ε, ε, αρχές να μπορούν να μπορούν να συνεργάζονται είτε σε δικαστικό είτε σε αστυνομικό επίπεδο και να χρησιμοποιηθούν ε, διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ξεπερνώντας ε, τα εμπόδια <clears throat> που αντιμετωπίζει κάθε χώρα να υπάρξει ένα Asset Recovery Office ε, να μην είναι μόνο βέβαια η μοναδική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά που θα μπορέσει, που θα δώσει την ικανότητα να συνδυάσουμε ε, διάφορες εθνικές τράπεζες δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε πού επενδύονται τα προϊόντα των δραστηριοτήτων αυτών της μαφίας και να μπορέσουμε να δούμε, ας πούμε, πού γίνονται οι επενδύσεις, ε, ε, πώς ξεπλένεται το χρήμα. Όλα αυτά βοηθάνε. Ευχαριστώ, εδώ, ε, ευχαριστώ. Σταματάω εδώ, Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας βέβαια και να συζητήσουμε και τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας. Κύριε Φάβα, ένα λεπτό. Απλώς να πω ότι ε, χαίρομαι ε, που βρίσκομαι εδώ, που, ξανά, που συναντάω ξανά τον πρόεδρο Μωράες. Ε, όλα τα είπε η κυρία Μπίντη και τόσο καλά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Απλώς Πιστεύω ότι τώρα χρειάζεται μια πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία από αυτήν του παρελθόντος και πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι διότι θα εκχωρείται και ένα μέρος της ε, ε, ε, κρατικής αρμοδιότητας, εξουσίας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μαφία έχει απλωθεί σε όλες τις χώρες. υπάρχει μια νέα οδηγία για την κατάσχεση και μια εισαγγελία η οποία θα ασχολείται όχι μόνο, με την, όχι μόνο με τις απάτες αλλά και με την αμαφία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα νομοθετικά προϊόντα τα οποία έχουμε παράγει. Ο κύριος Ούβα. Πρόεδρε, να σας πω ότι σαν Επιτροπή κατά της μαφίας δεν έχουμε απλώς ε, ε, συντάξει μία έκθεση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ε, όλους όσους κάνανε παρεμβάσεις. Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα βέβαια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μαφία εξελίσσεται και είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε να απαντήσω την κυρία Φεράρα όσον αφορά το, ε, ε, την υπηρεσία αυτή για την κατάσχεση των αγαθών. Χρειάζεται και χρήματα αλλά και ανθρώπινους πόρους. Δηλαδή ακόμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχουν γίνει απαραίτητοι διορισμοί για το προσωπικό. Ε, δεν θέλω να μπω τώρα ε, σε εσωτερικούς ε, πολέμους, αλλά τέλος πάντων να σας πω ότι προφανώς δεν υπάρχει κακή πίστη ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να επιταχύνουμε την, την, την αντίδρασή μας. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιταλία προσπαθεί να κάνει ένα πόλεμο ανάμεσα, ε, να κάνει ένα πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Κυρία Σκοπελίτη. Απλώς να χαιρετήσω τα μέλη της Επιτροπής και να τους ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον αλλά και για το γεγονός ότι θέλησαν να συμπεριλάβουν αυτό το σημείο της μαφίας στην ημερήσια διάταξη υπογραμμίζω και προσθέτω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Μπίντι και η κυρία Γκαραβίνη, την ανάγκη να δώσουμε αυτόν τον πόλεμο όλοι μαζί από κοινού. Διότι το πρόβλημα της μαφίας, το οποίο δημιουργήθηκε και ξεκίνησε βέβαια στην Ιταλία και μας δημιούργησε τέτοια τεράστια προβλήματα, είναι, ε, οδηγήθηκε στην κατάσταση αυτή διότι ακριβώς δεν θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να δούμε το πρόβλημα. Θα πρέπει η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι η μαφία δεν είναι ένα πρόβλημα της Νότιας Ιταλίας ή της Ιταλίας εν γέννη. Είναι ένα πρόβλημα τα οποία, το οποίο αφορά όλους μας. Η μαφία επενδύει και επενδύει πού, εκεί που υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Άρα θα πρέπει όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο όπου ε, θα έχουμε όλη την, ε, την δύναμη να πούμε όχι. Άρα είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Με τα όσα έγιναν, ας πούμε, πριν από λίγα χρόνια στη Γερμανία και θα πρέπει να εκφράσουμε όλοι μας ε, την θέληση να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο ενδεχόμενα να μην φαίνεται αλλά ακριβώς επειδή δεν φαίνεται είναι πιο ε, επικίνδυνο και ύπουλο. Νομίζω ότι έληξε ο χρόνος ε, που είχαμε στη διάθεσή μας και ζητώ συγγνώμη ε, από τα μέλη της ε, άλλης, τον, από τα, μέλη της Επιτροπής μας που τους ευχαριστώ για την παρουσία τους αλλά δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δικαστικούς αλλά και τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις εργασίες της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την προσοχή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίντι. Είναι κρίμα που πρέπει να κλείσουμε αυτή την εξαιρετική συζήτηση ε, που ήταν τόσο υψηλού επίπεδου. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο επίπεδο οριμότητας τώρα στη δουλειά που κάνετε και εσείς και εμείς. Πέρα από την Επιτροπή ΚΡΙΜ, μετά από αυτήν εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ εις ό,τι αφορά το θέμα των αξιόπινων πράξεων της εγκληματικότητας. Και εδώ Έχουμε και σε αυτή τη θητεία και στην προηγούμενη ε, και εξαιρετικούς συναδέλφους από την Ιταλία. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Ιταλικού Κοινοβουλίου, όσους μίλησαν και όσους δεν μίλησαν. Υπάρχει τώρα μακρά ιστορία ε, συνεργασίας μεταξύ μας που καταλήγει σε πρακτικό περιεχόμενο δουλειάς. Τώρα το πιο σημαντικό είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία για να κάνουμε πράγματα υπέρ των πολιτών μας στην Ιταλία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια συζήτηση, αυτή ήταν μια ε, συζήτηση σε βάθος ε, όπως είπε και η Κατερίνα Κινίτσι ε, και βέβαια ε, το πιο σημαντικό που τονίστηκε είναι η ανάγκη εφαρμογής νομοθεσίας. Ήταν πάρα πολύ καλό που κάναμε τη συζήτηση αυτή προς το τέλος της Ιταλικής Προεδρίας. Ήταν η καλύτερη χρονική στιγμή τώρα. Με μεγάλη χαρά σας είδαμε και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας. Γιατί ανεξάρτητα από τα πορίσματα της Επιτροπής, αυτό αυτό το θεματολόγιο θα συνεχιστεί και στο μέλλον και υποθέτω ότι θα σας δούμε πάλι αρκετά σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εσάς και, τον, ε, και τους συναδέλφους σας. Um, um, Συνάδελφοι, προχωρούμε αμέσως στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Περιμένουμε όμως μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό μέχρι να γίνει η ανασύνταξη εδώ της ομάδας. Um, λοιπόν, ας αρχίσουμε πάλι με το επόμενο θέμα, μελέτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στα χερσαία σύνορα και τα σημεία διέλευσης. 10 και 11 Νοεμβρίου ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μαζί με την Ιταλική Προεδρία ε, διοργάνωσαν ε, μια διάσκεψη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή τη χρονιά ήταν αφιερωμένη στο θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και μετανάστευση. Επίσης, ε, ο οργανισμός ολοκλήρωσε δύο μελέτες που υπέβαλε στην Επιτροπή. Αυτές εδώ. Η πρώτη εστιάζει στα θεμελιώδη δικαιώματα στα αεροδρόμια, η δεύτερη στα χερσαία σύνορα. Έχουμε εδώ τον κύριο Φρίσο Ρόσκαμ Άμπινγκ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας και Προσέγγισης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ήρθε για να κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Και μετά θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση και ερωτήσεις. Κύριε Άμπινγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΦΡΑ, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, να παρουσιάσει τις ε, πρόσφατες ε, εκθέσεις του που ε, άρχισαν σε αυτή τη διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έγινε στη Ρώμη πριν από δύο εβδομάδες και είχαμε τη χαρά να έχουμε και από την Αντιπρόεδρο Λότοβα πολύ σημαντική συμβολή. Τώρα θέλω εν συντομία να σας παρουσιάσω τις δύο εκθέσεις που δημοσιεύσαμε. Οι δύο εκθέσεις ε, ολοκληρώνουν μια τριλογία που άρχισε από πέρσι. Ε, είχαμε και ελέγχους στα θαλάσσια σύνορα που άρχισε στην ίδια Επιτροπή αυτό το Μάρτιο. Τώρα ολοκληρώνουμε την έρευνα και παρουσιάζουμε τα ευρήματά μας εις ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στα αεροδρόμια και στα σημεία διέλευσης χερσαίων συνόρων. Εξετάσαμε... τι κάναμε. Εξετάσαμε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται και στο κεκτημένο Σέγγεν που περιλαμβάνει και τον κώδικα συνόρων Σέγγεν όπως ξέρετε και βλέπουμε σε ποιο βαθμό γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και βασικές αρχές από τους συνοριοφύλακες. Κάναμε πολλές, ε, πήραμε συνεντεύξεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνοριοφύλακες ε, σε 11 κράτη-μέλη στο Μαρόκο, την Τουρκία, τη Σερβία, την Ουκρανία Κάναμε και μια έρευνα η οποία ε, συμπεριέλαβε 400 συνοριοφύλακες με πολύ χρήσιμα δεδομένα. Και όλο το πρόγραμμα συντονίστηκε ε, εκ του σύνεγγης από συναδέλφους της Frontex. Πρέπει να τονίσω ότι κυρίως είδαμε τους ελέγχους συνόρων σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών, όχι υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ, Διαπιστώσαμε ότι ε, οι έλεγχοι στα αεροδρόμια και στα χερσαία σύνορα γίνονται ως ρουτίνα, χωρίς επεισόδια. Κάποιες σοβαρές προκλήσεις παρόλα αυτά ε, πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ταξιδιωτών και σε πέντε τομείς εντοπίσαμε δυνατότητες βελτίωσης και έχουμε γνωμοδοτήσεις και συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Το πρώτο αφορά το σημαντικό θέμα ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Ε, τα πέντε σημεία θα σας τα παρουσιάσω. Το δεύτερο αφορά το θέμα της πρόσβασης στην πληροφόρηση και προσφυγή, ε, προσωρινή κυδαιμονία για παιδιά και ε, αντιπροσώπευση σε μη συνοδευόμενα, ε, ε, ιδιωτική ζωή και προστασία δεδομένων και προσωρινή κράτηση. Τώρα, βλέπουμε εδώ στην επόμενη διαφάνεια, εις ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, αυτό που είδαμε ως προκλησή είναι η σαφήνεια αυτού που σημαίνει ενδείξεις ε, μιας επιθυμίας για αίτηση για διεθνή προστασία. Σε κάποιες περιπτώσεις που θεωρούμε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός τους, αν κάποιος για παράδειγμα λέει ότι φοβούμε ότι θα με σκοτώσουν άμα επιστρέψω και δεν είμαι πολιτικός πρόσφυγας και ε, ζητώ άσυλο, ε, αυτό αν το έλεγε το πρώτο δεν ε, δίδεται συνέχεια όπως έπρεπε. Αυτομάτως τον παρέπεμπαν σε διαδικασίες ασύλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης ε, είδαμε, η έρευνα έδειξε, ότι οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες ε, δεν αντιμετωπίστηκαν ατομικά ε, ακόμα και αν υπήρχαν σαφείς ανάγκες για προστασία. Μπορέσαμε επίσης να δούμε κάποιες πρακτικές καλές, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά εξειδικευμένες ομάδες στο, και στο αεροδρόμιο και στα χερσαία σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Εκεί ε, είδαμε καλές ε, προϋπο... ε, συνθήκες ε, παραπομπής εκείνων που ήθελαν, χρειάζονταν διεθνή προστασία. Ο αριθμό τους ήταν σημαντικός τα τελευταία χρόνια. Εδώ δείχνει η διαφάνεια ότι όπως σας είπα, μόνο αν έλεγαν ξεκάθαρα είμαι πρόσφυγας, αυτό αναγνωρίζει το ότι θα έπρεπε να κινήσει διαδικασίες ασύλου. Ε, στις, περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις ε, δεν ε, έδιναν συνέχεια οι συνοριοφύλακες αν δεν ήταν ρητή η επιθυμία. 64% αντιδρούσαν στα χερσαία σύνορα σε αιτήματα που δεν ήταν σαφώς διατυπωμένα, δηλαδή είμαι πρόσφυγας, και 30% των αυτών που έδωσαν συνέντευξη είπαν σαφώς ότι δεν προέβαιναν σε, σε, λήψη μέτρων, σε ανάληψη δράσης. Ένα άλλο θέμα που μπορεί να βελτιωθεί και θέλουμε να σας το δείξουμε παρουσιάζει στην επόμενη διαφάνεια, δηλαδή πρόσβαση στην πληροφόρηση. Εδώ εντοπίζουμε τρεις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, συστηματική παροχή πληροφοριών σχετικά με το σκοπό και την διαδικασία κάποιων ελέγχων, ιδιαίτερα δεύτερης γραμμής ελέγχων μετά από έναν πρώτο έλεγχο όταν δηλαδή ε, οι αρχές των συνόρων θεωρούν ότι χρειάζεται δεύτερης γραμμής έλεγχος, σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι ο σκοπός και η διαδικασία δεν είχαν γνωστοποιηθεί επαρκώς. Αυτό όμως ο κώδικας Σέγγεν το προβλέπει στο άρθρο 7. Το ίδιο ισχύει όταν σε κάποιον ε, υπάρχει άρνηση εισόδου για κάποιον. Σε όλες τις περιπτώσεις ε, πρέπει να δίνονται ε, πληροφορίες σε σχέση με νομική ε, συνδρομή που πρέπει να αναζητηθεί. Τρίτον, αποτελεσματική πρόσβαση σε οργανώσεις που παρέχουν νομικές συμβουλές και διερμηνία. Αυτό υπάρχει σε όλα τα χερσαία σύνορα. Ε, προβλήματα γλωσσικά εντοπίστηκαν επίσης και τα οποία καταλαβαίνετε ότι ε, παρεμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ συνοριοφυλάκων και ενός ε, ε πολίτη από τρίτη χώρα. Λιγότεροι από τους μισούς από τους αξιωματικούς που εξετάσαμε και ρωτήσαμε στο αεροδρόμιο και στα χερσαία σύνορα είπαν ότι δίνουν πληροφορίες σε σχέση με το σκοπό και τη διαδικασία. Λιγότεροι από τους μισούς. Εις ό,τι αφορά την άρνηση εισόδου, η έρευνα έδειξε ότι πολλοί αξιωματικοί δεν δίνουν πληροφορίες σε σχέση με την νομική υποστήριξη. Αν, αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται όμως αν σας αρνηθούν την είσοδο. Τέλος, ε, πρόσβαση σε οργανώσεις που ε, δίνουν ε, υποστήριξη υπάρχουν Υπάρχει ο, η Πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες, η Επιτροπή ε, για την πρόληψη βασανιστήριων. Ε, είδαμε ότι στο Φιουμιτσίνο είναι καλή η πρακτική που ακολουθείται στη Ρώμη, όπου υπάρχει ένα γραφείο πληροφόρησης το οποίο ενημερώνει και παρέχει και διερμηνία σε ε, πολίτες τρίτων χωρών, ιδιαίτερα του άσυλο, αλλά και σε ταξιδιώτες που δεν γίνονται δεκτοί και δεν τους επιτρέπεται η στη χώρα. Πάμε στο τρίτο τομέα που ανησυχεί τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με βάση την έρευνα που έγινε, που αφορά την ε, ευάλωτη θέση μη συνοδευομένων παιδιών. Αυτό που είδαμε είναι ότι οι ρυθμίσεις δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές στις χώρες ε, που, όπου κάναμε την έρευνα κατά την ώρα του ελέγχου δεύτερης γραμμής όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενη παραπομπή. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό το στάδιο ένας ανεξάρτητος αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι παρόν για να διασφαλίσει ότι θα προστατευθούν τα συμφέροντα των παιδιών. Θα πρέπει να υπάρχει ένας προσωρινός ε, αντιπρόσωπος και δαιμόνας των παιδιών. Στο Σκύπολ του Άμστερνταμ είδαμε μια καλή πρακτική όπου όλα τα παιδιά πρώτα ε, μπαίνουν σε ένα χώρο υποδοχής ε, και εκεί ε, ο υπεύθυνο για αυτά τα συναντά και είναι παρόν όταν μιλήσουν με την αστυνομία. Το δεύτερο θέμα που μας απασχολεί είναι η ευαισθησία αυτή, η ευαλωτότητα των παιδιών. Ξέρουμε από την έρευνα των συνοριοφυλάκων ε, ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι για να χειρίζονται τα παιδιά. Και μας είπαν οι συνοριοφύλακες ότι θέλουν πολύ να εκπαιδευτούν καλύτερα για να αντιμετωπίζουν τα ευάλωτα παιδιά και τις ειδικέ τους ανάγκες. Εδώ έχουμε μια καλή πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ όπου κάναμε έρευνα, όπου εκεί ε, έχουμε αξιωματικούς ε, από το Τμήμα Μετανάστευσης ε, που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στα παιδιά και κάθε φυλάκιο συνόρων έχει κάποιον ειδικό στα παιδιά. Άλλο θέμα, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία δεδομένων. Εδώ διαπιστώνουμε ότι όλοι οι συνοριοφύλακες δεν ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για τις διαδικασίες ε, που πρέπει να ακολουθήσουν αν τους αρνηθούν την είσοδο. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και ποσοστό, μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων και στο σύστημα SIS και στο σύστημα VIS ε, ε, για το σύστημα πληροφόρησης Schengen και Visas. Και πολλές φορές οι συνοριοφύλακες λένε ότι ε, πράγματι οι βάσεις δεδομένων έχουν ε, υψηλό ποσοστό σφαλμάτων. Οπότε οποιαδήποτε θέση που στηρίζεται σε αυτή τη βάση δεδομένων επηρεάζει πάρα πολύ τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ε, το, η δεύτερη πρόκληση είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα επαγγελματικής διαρμηνίας έγκαιρα. Ρωτήσαμε τους αξιωματικούς εάν βοηθούνται από άλλους ταξιδιώτες αν κάποιος έχει πρόβλημα επικοινωνίας και η πλειοψηφία 100 αξιωματικών στα πέντε αεροδρόμια που πήγαμε και θα το δείξουμε στην επόμενη διαφάνεια αυτό δηλαδή 67% κατά μέσον όρο, στηρίζονται και ε, στη βοήθεια άλλων ταξιδιωτών που θα βοηθήσουν στη διαρμηνία. Και αυτό βεβαίω έχει ε, επιπτώσει όχι μόνο στην ποιότητα τη επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένη και συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού αναγκών ε, υποστήριξη, αλλά επηρεάζει και την προστασία δεδομένων. Αυτό είναι προβληματικό γιατί ε, οι συνοριοφύλακες δεν ε, ε, γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα προστασίας δεδομένων. 45% των εργαζομένων στα αεροδρόμια είπαν ότι είχαν εκπαίδευση και 34% στα χερσαία σύνορα. Πέμπτο και τελευταίο μέλημά μας, οι συνθήκες κατά την προσωρινή κράτηση. Φαίνεται ότι είναι πρόκληση αυτό το θέμα, μια δυσκολία σε πολλά χερσαία σύνορα, σε σημεία διέλευση δηλαδή χερσαίων σύνορων. Διαθεσιμότητα τροφίμων και νερού, πρόσβαση σε τουαλέτες, ε, χώρος για ε, κάποια ξεκούραση ε, πριν από άλλον έλεγχο ή επιστροφή. Θεραπεία, ε, ε, μεταχείριση ευάλωτων προσώπων σε χώρους κράτησης, σε ε, υπήρχαν αναφορέ ότι δεν, έκλειναν, δεν κλείδωναν οι τουαλέτες ε, όταν έπρεπε να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο. Ε, τέλος, η επικοινωνία με τον εξωκόσμο πολλές φορές δεν είχαν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους. εδώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ε, εξουσιοδοτήσουν κάποιον, να επικοινωνήσει. Ε, εδώ στο Μάντσεστερ έχουμε πολύ, ε, πολλά υποσχόμενες πρακτικές. Τους δίνουν κινητά για να βάλουν την κάρτα SIM και να έχουν έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης και στην επικοινωνία και να μιλήσουν με ανθρώπους που θα τους εφοδιάσουν με απαραίτητα έγγραφα ενδεχομένως να τους βοηθήσουν. Τέλος, ε, το follow-up, η συνέχιση που ε, κάνει, θέλει να κάνει ο οργανισμός μας, ε, με τη Frontex καταρχήν. Εδώ σκεπτόμαστε να συνεργαστούμε μαζί τους ε, για να καταρτήσουμε ένα εγχειρίδιο για τα παιδιά. Εκείνοι το έχουν ετοιμάσει. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με άλλους οργανισμούς ε, τη Europol, την Σέπολ. Ε, Θέλουμε να τους εντάξουμε σε ένα πρακτικό follow-up και να δούμε ποιες συστάσεις ενδεχομένως θα ε, προωθήσουμε για να εφαρμόζονται και από εκείνους. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην αξιολόγηση ε, στο Σένιεν και του χρόνου θα αρχίσουμε ένα σημαντικό έργο πάνω στα βιομετρικά δεδομένα που θα δούμε τα στοιχεία θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με τις βιομετρικές μεθόδους ε, ε, αναγνώρισης ταυτότητας, ταυτοποίησης. Αυτά ήθελα να σας πω. Και για να κλείσω, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα συμπεράσματα που είναι πολύ εκτενή από τη διάσκεψη και ελπίζω να μπορέσουμε να τα διανύμουμε στην Επιτροπή σας κάποια στιγμή αργότερα γιατί αφορούν μεταξύ άλλων το θέμα των ελέγχων των συνόρων και μια προσέγγιση που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και αφορά και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Αυτά τα είπαμε στην διάσκεψη που είχαμε 300 εκπροσώπους από ε, διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς, μη κυβερνητικ... κυβερνητικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές και ε, θα ήθελα πραγματικά να σας πω ότι αξίζει να διαβάσετε τα συμπεράσματα της διάσκεψης. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση, τι δύο εκθέσεις. Η Κομισιόν, η Frontex επιθυμεί να... Η Κομισιόν θέλει να κάνει κάποια σχόλια, όχι. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι. Η Frontex... Ένα σύντομο σχόλιο από τη Frontex. Ευχαριστώ. Είμαι υπεύθυνη από τη Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ ε, τον οργανισμό ΦΡΑ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την πολύ αυτή στέρεη έρευνα η οποία συμπληρώνει την περσινή έκθεση για τα θαλάσσια σύνορα και τα εξωτερικά σύνορα. Εμείς μελετήσαμε πολύ προσεκτικά την έκθεση αυτή και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβω με θέματα που μας αφορούν στις επιχειρήσεις μας και το ίδιο θα κάνουμε και με τούτες τις εκθέσεις για τα αεροδρόμια και τα χερσαία σύνορα μετά τη δημοσίευσή τους. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι σε κάποια σημεία διέλευσης δεν κινητοποιεί το μηχανισμός παραπομπής όταν υπάρχουν ευάλωτα πρόσωπα ή όταν χρειάζονται διεθνή προστασία, αλλά γενικά εμείς σημειώνουμε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό που το έχουμε συζητήσει ε, της έλλειψης δικτών φιλικών προς τους χρήστες για τη διεθνή προστασία και τα ευάλωτα πρόσωπα και θέλουμε προληπτικά μέτρα περισσότερα από την πλευρά των συνοριοφυλάκων, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί παραπομπής. Αρχίσαμε συζητήσεις ε, και με το δικό σας το γραφείο και την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες για να καταρτήσουμε μοντέλο κατάρτισης εκπαίδευσης πάνω σε ένα ε, ε, σχέδιο ε, αντιμετώπισης προσφύγων που θα καλύπτει ετούντες άσυλο στα σύνορα. Επίσης είναι ευπρόσδεκτη η ιδέα να ε, δοθούν τα εγχειρίδια για να εντοπίζονται παιδιά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο στα σύνορα και τώρα θα γίνει αυτό και στα αεροδρόμια. Επίσης σημειώνουμε την κατεπίγουσα ανάγκη να δώσουμε το εγχειρίδιο αυτό και στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα. Εμείς ολοκληρώσαμε μια κοινή επιχείρηση πρόσφατα ε, σε σχέση με αυτό το εγχειρίδιο, δηλαδή τα, ε, ε, εντοπισμός παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο, ήταν μια κοινή επιχείρηση πολύ ειδική, γιατί ήταν σε συνεργασία με ειδικού στην αντιμετώπιση παιδιών. Είχε μεγάλη επιτυχία, ήταν μια επιτυχή σύμπραξη που αποτελεί μοντέλο και για μελλοντικές συνεργασίες ε, που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα σε ευαίσθητους τομείς. Ε, επίσης η εκπαίδευση συνεχίζεται στα θέματα που θέσατε και την ανάγκη να εξυγχρονίσουμε περισσότερο το θέμα προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Frontex, να μην εστιάσουμε μόνο στα, ε, στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση παιδιών ή προσφύγων κλπ, αλλά να έχουμε εκπαίδευση ε, συνολικότερη σε ό,τι αφορά το προφίλ των συνοριοφυλάκων σε όλα τα σύνορα. Ε, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι τις συστάσεις σας τις ε, εξετάζουμε πολύ προσεκτικά και θα προσπαθήσουμε την υποστήριξή σας να τις εφαρμόσουμε. Ωραία. Αυτές οι μελέτες αντικατοπτρίζουν πάρα πολύ δουλειά που έχει γίνει για τον έλεγχο των λιμένων και των αεροδρομίων. Γνωρί... Πολλοί συνάδελφοι ξέρουν ε, περιπτώσεις ε, ανθρώπων που συνελήφθησαν ε, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, που στερήθηκαν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Αυτά είναι οι πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Δημιουργώντας αυτές τις δύο μελέτες, οφείλω να ομολογήσω ότι το έργο σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και κανείς το έχει κάνει στο παρελθόν. Καταρχάς, επομένω σας συγχαίρω που το κάνετε. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που ζητάνε το λόγο και ε, τα θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στέρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων εσείς έχετε καλύψει τη σύμβαση και τον χάρτη θεμελιωδών, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είπατε τι συμβαίνει στα αεροδρόμια. Ίσως κάποια μέλη εδώ, κάποιοι συνάδελφοι έχουν, ήταν, έχουν, έχουν ε, παρευρεθεί, υπήρξαν μάρτυρες τέτοιου είδους ε, περιστάσεων, περιστατικών. Υπάρχουν προφανώς και κάποια, κάποιες δυνατότητες που προσφέρονται σε, εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγγνώμη. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ε, κάποια νομοθεσία κατά των διακρίσεων που θα προστατεύσει τα άτομα στους ελέγχους, στα σύνορα ή στα αεροδρόμια. Υπάρχει κάποιες, υπάρχουν κάποιες διατάξεις στη μεταναστευτική πολιτική, στην νομοθεσία που αφορά την, τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα επέτρεπε αυτού του είδους τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται με καλύτερο τρόπο. Ξέρω, ας πούμε, ότι πάρα πολλές φορές η εθνική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια γιατί θεωρούμε ότι είναι μια ζώνη όπου ο καθένας μπορεί να κάνει θέλει. Γιατί τα λέω, ότι όταν κάποιος σε συλλαμβάνει, όταν σε σταματάνε και σε ψάχνουν, πολλά μπορούν να συμβούν και είχα την ευκαιρία να εξετάσω αυτές τις ε, εκθέσεις και μιλάτε για τη σύμβαση, μιλάτε για τον, για τον χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Η πραγματικότητα όμως του να σε σταματήσουν σε ένα λιμάνι, σε ένα αεροδρόμιο, να σε ψάξουν, να σε γδίσουν για να σε ψάξουν ε, και να, σε, να βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο το θέμα. Και ε, ρωτώ, έχετε εξετάσει τις εθνικές νομοθεσίες. Στην Πολωνία πρόσφατα ένας ένας σε έναν ζητήσανε να βγάζει συνέχεια το τουρμπάνι του ε, μπορούσαν να το ε, τσεκάρουν, να το ελέγξουν αλλά παρόλα αυτά συνέχισαν να το ζητάνε να το βγάλει για να τον ε, για να καταρακώσουν την αξιοπρέπεια ε, τελικά κατέληξε στο δικαστήριο η ιστορία αυτή αλλά τέλος πάντων ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η έκθεση σας ε, ή και η μελέτη σας είναι εξαιρετική, αλλά υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα. Είναι πάρα πολύ ε, εφικτό να, ε, κάποιος να ταπεινώσει κάποιον σε, στο, σε ένα αεροδρόμιο, σε σε ένα λιμάνι. Είναι δύσκολη η περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος κρατείται στο λιμάνι στο... και σε ένα αεροδρόμιο. Δεν λέω και σε, άλλες περι... Ε, ε, σε άλλους χώρους, αλλά εκεί συγκεκριμένα. Ο κύριος Κίρκοφ, Τίμωθη, έχει το λόγο. Είναι ενδιαφέρον και αυτό που αναφέρατε και πάνω σε αυτό. Ε, θέλω και εγώ να κάνω κάποια σχόλια, αλλά από την άλλη πλευρά, διότι φυσικά η δουλειά των ε, αρχών επιβολής της νομοθεσίας ε, ή ε, των ανθρώπων που εργάζονται στα σύνορα. Έχουν τα καθήκοντά τους. Το αεροδρόμιο που ήταν αντικείμενο της μελέτης είναι το μεγαλύτερο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σίγουρα δέχεται πολλούς στην στην Ένωση, στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει ένα κενό εδώ, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Στην έκθεση Λέω ότι οι συνοριοφύλακες μπορεί να είναι έως και εχθρικοί ε, στην προφορική τους ε, επικοινωνία. Είναι όμως και θέμα προσωπικό. Εγώ έχω λάβει γνώση πολλών περιπτώσεων που αργότερα στο πλαίσιο μιας νομικής διαδικασίας υποστήριξαν ορισμένοι ότι δεν τους φέρθηκαν με αρμόζοντα τρόπο οι συνοριοφύλακες. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν κατάλαβαν καλά ή ότι οι συγκεκριμένοι αυτοί άνθρωποι ε, ισχυρίστηκαν την έλλειψη φιλικής συμπεριφοράς, ας πούμε, ε, ή εχθρικής στάσης ε, ως επιχείρημα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι όμως δυνατόν ε, να λάβουμε υπόψη, μάλλον πρέπει να λάβουμε υπόψη στο γεγονό ότι κάποιος πρέπει πρώτα να γίνει δεκτός από την ε, δικαιοδοτική αρχή της χώρας. Στο αεροδρόμιο δεν ισχύει αυτό. Εκεί δεν καλύπτεται νομικά ο εν λόγω ε, πολίτης που έρχεται. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Βέβαια εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει το ζήτημα εισδοχή σε μια χώρα. Με βάση τους κανόνες της χώρας. Έχουμε βέβαια τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το θέμα. Ναι, μεν καλωσορίζω την έκθεση και το έργο που έχει γίνει, αλλά θεωρώ ότι σε κάποιο μέρος του είναι ανεδαφικό, σε κάποιο βαθμό προτείνει κάποια επίπεδα σεβασμού τα οποία νομίζω και φοβούμε ότι στον κόσμο που ζούμε πολύ δύσκολα να τα εγγυηθεί κανείς. Τα πρότυπα ε, της, ε, των αεροδρομίων του Ηνωμένου Βασιλού είναι ε, υψηλά, έχουμε ελέγχους για να βλέπουμε πώς μεταχειρίζονται οι συνοδεύτες τα παιδιά, ιδίω. το ξέρει και ο Κλοντ, δεν είναι παντού τα πρότυπά μας τέλεια, πρέπει να βελτιωθούν. Όμως, όπως είπα, οι αρμοδιότητες και τα νομικά αποτελέσματα όπως προβάλλονται στην έκθεση. Νομίζω ότι χαρακτηρίζονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένα πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Πρόεδρος, πρέπει να υπάρχει και ένα νόμιμο, ε, συγγνώμη, και ένα ασφαλής νομικό περιβάλλον στα αεροδρόμια. σε λιμάνια και αεροδρόμια. Αυτό είναι σημαντικό σίγουρα. Την άλλη πλευρά, η συνέπεια που πρέπει να υπάρχει και συνεκτικότητα στις μεταχείρισεις στα αεροδρόμια και στους λιμένες. Χωρίς να θα στοχοποιήσω την Πολωνία. Ε, έγινε όμως κάτι εκεί που δεν έγινε στη Γερμανία για παράδειγμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται λοιπόν, ποια είναι η συμπεριφορά στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και η εμπειρία μου ε, διδάσκει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές πρακτικές ε, στα αεροδρόμια για στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα θέμα ακόμη που πρέπει πιστεύω να θέσουμε. Το επόμενο ερώτημα είναι από την Birgit Ζίπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα καταρχάς να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τα αποτελέσματα της διάσκεψης ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μιλήσατε για την ε, προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα για την καταπολέμηση τη παράνομη διακίνηση. Ένα σύντομο σχόλιο ήταν αυτό εν παρόδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά του νοριακού ελέγχου και ποιε είναι οι προκλήσει που αναφέρετε στην ε, έκθεσή σα. Έχω την εξή ερώτηση. Γιατί όταν έχουμε το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν ε, κατάλληλες αίθουσες, ε, δεν ε, υπάρχει η γλωσσική υποστήριξη, δεν υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση για τα παιδιά και άλλες ομάδες ευάλωτες κτλ. Ποιος φταίει, δεν το γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές που πρέπει να λάβουν το καθήκον. Δεν υπάρχει προθυμία να δαπανηθούν πόροι για εξειδικευμένο προσωπικό για όλα αυτά τα θέματα και ένα άλλο ερώτημα. Τελικά, οι αρμόδιες αρχές είναι πρόθυμες και διατεθειμένες να αλλάξουν ε, την οργανωτική δομή ή τα οικονομική, την οικονομική δομή για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις. Πρόεδρος, ωραία ερώτηση. Ο Χουάν Φερνάντο είναι τώρα επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στην ίδια γραμμή και θα εκφράσω και εγώ τις ίδιες ανησυχίες μας προλέσσαντες συναδέλφους μου. Φυσικά και όλοι αναγνωρίζουμε το ρόλο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την ανάλυση και την παροχή ε, πληροφοριών διεξοδικών για το τι συμβαίνει στα σύνορα, στα αεροδρόμια και στα λιμάνια και τα θέματα τα οποία τις προκλήσεις. Βέβαια, Γνωρίζουμε όλοι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνιακό. Είναι προφανές ότι τα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι πολλοί από αυτούς τέλο πάντων σε ε, κάθε, κάθε εβδομάδα ή εμείς οι ευρωβουλευτές σχεδόν καθημερινά ζουν αυτές τις εμπειρίες, αυτούς τους ε, συνοριακούς ελέγχους που δημιουργούν ανησυχίες ε, σε ό,τι αφορά τα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατάρτιση υπάρχει, εκπαίδευση, κάποια που εμείς έχουμε και νομική, ε, νομικό υπόβαθρο, ξέρουμε τι περίπτωση πρόκειται, αλλά εκατομμύρια άλλοι συμπολίτε μα δεν έχουν ιδέα για το ποια είναι τα νομικά πρότυπα και οι κανόνες που δικαιολογούν τέτοιου είδους συμπεριφορές στα αεροδρόμια. Δεν γνωρίζουν κατά πόσον υπάρχει αυτό το λεγόμενο profiling που συνιστά διακριτική μεταχείριση. Δηλαδή ότι στοχοθετούνται, ουσιαστικά στοχοποιούνται κάποιοι ε, συγκεκριμένοι άνθρωποι και ελέγχονται πιο συχνά από άλλους ούτε γνωρίζουν αν έχουν ε, δυνατότητες, κάποιο ενδικό μέσο που να χρησιμοποιήσουν κτλ. Επομένως, ερώτηση, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για να τα καταφέρουν καλύτερα στον τομέα αυτό. Δηλαδή, να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη και να τους πούμε ότι ξέρετε υπάρχει ο χάρτης των δικαιωμάτων. Που ε, μπορεί να παίξει ένα ρόλο εδώ. Εμείς λοιπόν, ε, νομοθέτες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να έχουμε έναν συνεκτικό νομικό κανόνα, ώστε οι εθνικοί κανόνες και ρυθμίσεις να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και να έχουν μια νομική δεσμευτική ισχύ. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση, την επιχειρησιακή των ε, σχεδίων ασφαλείας γνωρίζουν ότι υπάρχουν ζητήματα που άπτονται ε, της των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Διότι εμείς, οποιοςδήποτε άλλος θα προσάρει, να στάσεις μας να εμείς λέω, Έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη. Ε, προσλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι όμως ε, για τους ελέγχους αυτούς που δεν έχουν ιδέα και που το μόνο που κάνουν να ακολουθούν εντολές. Και όταν τολμήσει κανείς να θέσει ένα νομικό ζήτημα, σεβασμός ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που είναι θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρώνεται στο χάρτη Μα λένε τότε αυτοί λοιπόν, όταν το θέτουμε αυτό το ζήτημα, ακολουθούμε εντολέ και θα κάνετε ό,τι σα λέμε ακριβώ. Και θα κάνετε ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Θα υπακούσετε. Θα κάτσετε εδώ, δεν θα κουμπίσετε τι αποσκευέ σα. Θα σα ε, ψηλαφίσουμε κτλ. Πώ, Πώς θα φτάσουμε σε αυτή την πτυχή, σε αυτή την ψηλοποίηση και να κάνουμε τη διαφορά ψηλοποίηση όλων αυτών των κανόνων. Υπάρχουν ε, μελέτες, αναλύσεις. Πραγματικά είναι θετικές, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την... που μας είπες και για την εμπειρία σου στον JFK. στα αεροδρομία Το περιέγραψες πολύ παραστατικά. Je vous remercie. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ διαφωτιστικές ε, οι εκθέσεις για μια άγνωστη πτυχή του ελέγχου των πιστερικών συνόρων πιο συχνά τονίζουμε την πτυχή της ασφάλειας ε, και πολύ λιγότερο το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων. Και με τις εκθέσεις αυτές βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πιθανότητες προσφυγής, ε, ε, έχουμε κινδύνους διακριτικής μεταχείρισης, ιδίως ό,τι αφορά τα παιδιά. Πολύτιμες οι πληροφορίες. Τώρα λοιπόν πρέπει να τις μεταφράσουμε σε πράξεις. Τα κράτη-μέλη, κομισιόν, πώς υποδέχθηκαν τις προτάσεις δεν έχουν δεσμευτεί ήδη να εφαρμόσουν ορισμένε εξ αυτών. Ο Οργανισμό των Μελετών Δικαιωμάτων θα παρακολουθήσει την ελαιοποίηση των συστάσεων αυτών, ιδίω ε, με στόχο τα θεμελιώδη δικαιώματα να ε, ενταχθούν πιο πολύ ε, στην εφαρμογή των κανόνων Σέγγεν και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε εμείς στη νομοθετική μας δράση να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα αυτών των δύο εκθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Ο, ε, κυρία Σουίνμπερκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ναι, βλέπω ότι αντιμετωπίζετε πολλές προκλήσεις. τα συστήματα VIS, SIS, Eurodac, ανταλλαγή πληροφοριών τα χρησιμοποιούμε πολύ. Και μας ε, απασχολεί το πώς η Frontex κάνει τους ελέγχους ε, τηρώντας τους κανονισμούς του Δουβλίνου. Οι κανονισμοί του Δουβλίνου πώς ε, εφαρμόζονται, τηρούνται στα διάφορα κράτη-μέλη. το έχετε δει αυτό, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε και πάλι για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση των δύο εκθέσεων. Um, Αρχίζω με την ερώτησή σας σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας κυρίως στα σημεία διέλευση ετσαίων συνόρων και πώς ε, έχει να κάνει αυτό με το εθνικό δίκαιο. Δεν έχουμε κάνει ειδική έρευνα, αλλά ο κώδικας συνόρων Σέγγεν, που είναι ενωσιακή νομοθεσία και μέρος του κεκτημένου του Σέγγεν, εφαρμόζεται στους ελέγχους, ε, ώστε οι ταξιδιώτες να αντιμετωπίζονται ε, με αξιοπρέπεια να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά τους. Αυτό δεν είναι πέραν αμφιβολίας. Αυτό που κοιτάξαμε κυρίως στην έρευνά μας είναι το εξής, ότι όταν κρατούνται κάποιοι άνθρωποι και στερούνται την ελευθερία τους, θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνονται σχετικά με το τι θα γίνει, γιατί γίνεται και να τους προσφέρεται πρόσβαση επίσης σε νομική αρρωγή και να δίνεται σχετική πληροφόρηση. Εκεί διαπιστώνουμε ότι σίγουρα σε όλες τις περιπτώσεις δεν γίνεται σωστά, δεν δίνεται σωστά αυτή η πληροφόρηση. Τώρα το άλλο, το εθνικό profiling, η ταυτοποίηση ορισμένων ανθρώπων. Ε, αυτό που ρωτήσαμε τους συνοριοφύλακες και είπα ότι 400 συμμετείχαν, που είναι καλό δείγμα, και αυτό είναι παράρτημα στην έκθεσή μας και αξίζει να δείτε τις ερωτήσεις που τους κάναμε έτσι στα γρήγορα γιατί τους ρωτήσαμε σχετικά με το πώς κάνουν το profiling. Και είδαμε ότι γενικά ε, δεν υπάρχει συστηματική διακριτική μεταχείριση. Ε, υπήρχε όμως ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση και οι ταξιδιώτες που τους ρωτήσαμε είπαν ότι στο, στους ελέγχους δεύτερης γραμμής αντιμετωπίστηκαν με διακρίσεις. Το θέμα του profiling για συγκεκριμένες ε, χώρες ε, έχουμε ε, δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο το οποίο πάλι αφορούσε την ομάδα στόχο των ανθρώπων που εφαρμόζουν το profiling. Καλό είναι λοιπόν να λαμβάνετε υπόψη, μπορούν να το λαμβάνουν υπόψη και κάναμε συστάσεις και στους συναδέλφους από τη Frontex να το χρησιμοποιούν όσο γίνεται περισσότερο και να το χρησιμοποιούν και στη, στα προγράμματα κατάρτισης που κάνουν. Η ερώτηση του κυρίου Κέρκοπ. Θέλω να πω ότι Πήγαμε στο Μάντσεστερ γιατί καταρχήν σκεφτήκαμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, του Heathrow. Αλλά δεν είχαμε πρόσβαση στο τέλος του Heathrow. Δεν, μπορούσαμε ε, να κάνουμε την έρευνα εκεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο στο, πήγαμε στο Μάντσεστερ λοιπόν και είναι και σχετικά μεγάλο αεροδρόμιο και μπορέσαμε να ε, εξετάσουμε τα σημεία που θέλαμε. Να πω ότι στην περίληψη της έκθεσης για τα χερσαία σύνορα λέμε ότι τα, οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται με, με τρόπο που σέβεται την, ε, ε, ε, ε τους ταξιδιώτες αν και πολλές φορές δεν χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη γλώσσα μπορεί κανείς να πει ότι πολλές φορές οφείλονται αυτά σε γλωσσικά εμπόδια. Είδαμε και πολύ θετικά παραδείγματα συμπεριφοράς συνοριοφυλάκων που ξεπερνούσαν την εντολή που είχαν. Η συνάδελφος που πήγε στο Φιουμιτσίνο σημείωσε ότι κάποιοι συνοριοφύλακες εκεί ε, αγόρασαν με δικά τους χρήματα νερό για τους κρατουμένους κάτω από δυσχερείς συνθήκες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει γενικά αρνητική στάση. Βέβαια θα πρέπει να ε, υπάρχει σεβασμό στην επικοινωνία και να γίνεται σωστή μεταχείριση ευάλωτων ανθρώπων. Η κυρία Σίπουλ ρωτάει γιατί δεν είναι περισσότερο γνωστά τα δικαιώματα που ε, ε, υπάρχουν και γιατί και, αν υπάρχει ε, προθυμία για να βελτιωθεί η κατάσταση και να υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα του κώδικα του Σέγγεν για παράδειγμα. Οι διατάξεις είναι σαφείς. Αυτό που σημειώσαμε και γι' αυτό παρέπεμψα στο παράρτημα με τις ερωτήσεις στους ενιοριοφύλακες είναι ότι όταν τους ρωτάμε ενδιαφέρεστε, θέλετε να εκπαιδευτείτε περισσότερο και αναφέρετε τους τομείς κατάρτισης που θέλετε ε, να συμμετέχετε. Είχαμε πολύ θετικές, πολλές θετικές απαντήσεις. Γιατί ο συνοριοφύλακα είπε: Δεν ξέρω πολλά για τα δικαιώματα των παιδιών ή για την προστασία των δεδομένων. Θέλω όμως να μάθω περισσότερα μέσα από κατάρτιση. Τώρα, σε ποιο βαθμό οι αρχές είναι πρόθυμες να επενδύσουν περισσότερα χρήματα για πρόσθετη κατάρτιση. Ε, δεν το ξέρω αυτό. Ελπίζω να είναι πρόθυμες. Αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί και με τους συναδέλφους από την ΣΕΠΟΛ, την ε, ε, Αστυνομική Ακαδημία και την ΕΑΣΟ και τη, με τη Frontex. Γιατί όλα αυτά ενδεχομένως ανάγονται στη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση από την πλευρά και των συνοριοφυλάκων και όχι μόνο από την πλευρά των ευάλωτων ανθρώπων που πρέπει να ξέρουν τα δικαιώματά τους. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίζουν ανθρώπους οι συνοριοφύλακες που είναι σε δυσχερή θέση. Ο κύριος ε, Γιάρα έχετε δίκιο βέβαια ε, υπάρχει χαμηλό επίπεδο ε, γνώσης ε, των δικαιωμάτων τους από ευάλωτα άτομα. Αυτό φαίνεται, φάνηκε από το 2008 που έγινε μεγάλη μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων. Ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Θα απαντήσω αναφέροντας δύο πρακτικά ζητήματα. Καταρχήν, η ΦΡΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οργανισμός δημοσιεύει όλο και περισσότερα εγχειρίδια ε, για τους ε, υπεύθυνου. Ε, αυτά είναι τα καλύτερα προϊόντα μας, παρόλο που διανέμονται δωρεάν. Δίνουν τη δυνατότητα για εκπαίδευση και για τους νομικούς, τους δικηγόρους που υπερασπίζονται ευάλωτα πρόσωπα και οι αρχές ενημερώνονται και για το ε, εθνικό profiling και για διάφορα θέματα που αφορούν προστασία δεδομένων, νόμο για τους πρόσφυγες, δίκαιο για τους πρόσφυγες. Αυτά τα εγχειρίδια δηλαδή καλύπτουν υπάρχουσες ανάγκες. Επίσης, αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχουν πολλές, πολλά υποσχόμενες πρακτικές, οι βέλτιστες πρακτικές αν θέλετε. Επίσης βλέπουμε ότι άλλα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτές οι καλές πρακτικές, αυτό που είπατε εσείς για την ε, ομοιομορφία πρακτικών στα διάφορα αεροδρόμια. Ελπίζομαι και είναι εύκολο να διασφαλίσουμε και αυτό το, ε, σε αυτό συμβάλλει η ΦΡΑ, ε, είναι να διαδοθούν αυτές οι πολλά υποσχόμενες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών. Ας πούμε, εγκλήματα μίσους. Τι κάναμε. Έχουμε μια ομάδα εργασίας για τα κράτη-μέλη, όπου διαδίδομαι, συζητούμε πρακτικές που φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα ήδη σε κάποιες χώρες. Η κυρία Ρεβοντελόν, εμείς συμβάλλουμε στις αξιολογήσεις του Σέγγεν αυτή είναι μια διαδικασία όπου όλο και περισσότερο ο οργανισμός μας, ε, ο ΦΡΑ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, καλείται να αποφανθεί. Αυτή είναι θετική εξέλιξη και στην Επιτροπή Αξιολόγηση Σέγγεν, όπου κληθήκαμε και εμείς να, δώσουμε μια, να κάνουμε μια αξιολόγηση για τη δομή των αξιολογήσεων Σέγγεν και πώς πρέπει να μετρούμε τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην αξιολόγηση κάποιων κρατών μελών που υπόκεινται σε αξιολογήσει Σέγγεν. Σε ό,τι αφορά την την τελευταία ερώτηση για τον κανονισμό Δουβλίνου, δεν έχω πολλά να πω τώρα, γιατί αυτή η συγκεκριμένη έρευνα δεν εξέτασε αυτή την παράμετρο. Δεν θέλω λοιπόν να προδικάσω άλλες μελέτες, ούτε να πω πράγματα τα οποία δεν στηρίζονται από τα απορίσματα αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο είπα στην αρχή. Να σας ευχαριστήσω όχι σας μόνο προσωπικά αλλά και όλη την ομάδα σας από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Διότι πρόκειται είναι ένα άκρος πολύπλοκο έργο. Λιμάνια και αεροδρόμια είναι άκρος νεφελώδης τομέα θα έλεγα, για να δει κανείς τα θέματα του profiling, της αξιοπρέπειας και εδώ γκρίζα νομική ζώνη. Δύσκολο το εγχείρημα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Και πραγματικά και από τα ερωτήματα των συναδέλφων θα διαπιστώσετε πόσο ήταν σημαντικό για μας που ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που μπήκε στην ημερήσια διάταξη και έγινε ε, μια τέτοια έκθεση. Είναι πολλά τα σημεία που θα μπορέσουμε να προωθήσουμε σε ό,τι αφορά τους κανόνες του Σέγγεν και άλλους κανόνες δεν είμαι πεπισμένος ότι καλύπτει παρκώς ε, τους πολίτες μας, τους προστατεύει παρκώς στα λιμάνια και στα αεροδρόμια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πιο ήπιοι με τα θέματα της ασφάλειας και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα αεροδρομία και τα άλλα. Αλλά τα θέματα της προστασίας, ε, της νομικής, ε, των ε, πιο ευάλωτων είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν ένιωσα έτσι και τόσο αισιόδοξο με αυτά που διάβασα στην έκθεση και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη στην Επιτροπή μας. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πτώση στο θέμα της ασφάλειας αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και συνεκτικότητα των κανόνων που ισχύουν στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Α, από ό,τι είδα έχουμε και μια ψηφοφορία στις 12 και 4. Επειδή όμως ε, πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, ίσως να γίνει και νωρίτερα η ψηφοφορία, πριν τις 12 και 4. Έτσι όπως πηγαίνουμε τουλάχιστον. Μήπως πρέπει να ενημερώσετε συναδέλφους ε, να έρθουν λίγο νωρίτερα. Αλλιώς θα περιμένουμε βέβαια μέχρι τις 12 και 4. Εντάξει, 12 και 4 γιατί είδα να γουρλώνετε τα μάτια και να κάνετε άλλες κινήσεις και χειρονομίες. Οκ, okay, αφήνω για τις 12 και 4 την ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω, όπως προβλεπόταν, η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 και 4. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκτης εξαμηνίας έκθεσης για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Στις 27 Νοεμβρίου η Επιτροπή ενέκρινε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 ε, τακτικό check-up της λειτουργίας ε, του χώρου του Σέγγεν, όπως το αποκαλούμε. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί, να έχουμε ένα στιγμιότυπο έτσι της κατάστασης και ελπίζω αυτό να αποτελέσει και τη φάση συζήτησης για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν, όπως ε, ήθιστε. Καλύπτει η έκθεση όλους τους τομείς του κεκτημένου του Σέγγεν, ιδίω διαχείριση εξωτερικών συνόρων, κατάργηση συνοριακών ελέγχων στα σφαιρικά σύνορα, και η περίοδος που καλύφθηκε την ε, τελευταία φορά ήταν η περίοδος από 1η Μαΐου 30 Οκτωβρίου 2014. Κάποια βασικά στοιχεία για να είμαι σύντομο στην παρουσίασή μου. Αν δει κανείς την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα, δεν εκπλήσεται που το βασικό πρόβλημα είναι η μαζική εισρωή, για να μην πω εισρωή ρεκόρ εισόδου, ιδίω στα νότια θαλάσσια σύνορα, Ιταλία πρώτα και Ελλάδα κατά δεύτερον. Αν δει τώρα τα ανατολικά χερσαία σύνορα, εκεί είναι σχετικά ήρεμη κατάσταση, η κρίση στην Ουκρανία. Θα να πω ότι δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε σημαντικές πιέσεις στα ανατολικά κράτη-μέλη, αλλά ίσως αυτή η κατάσταση αλλάξει πολύ γρήγορα. Ένα τελευταίο θέμα που τονίσαμε σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα ήταν και η συζήτηση που είχαμε τους τελευταίους μήνες για το πώς μπορούν οι συνοριακοί έλεγχοι ε, να συνεισφέρουν ε, στην ε, περίπτωση εντοπισμού των αποκαλούμενων ξένων μαχητών που πηγαίνουν στη Συρία και συμμετέχουν εκεί και επιστρέφουν ριζοσπαστικοποιημένοι πολλές φορές. Φυσικά απαιτούνται πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου ε, με τους νεαρκούς ελέγχους ε, δεν ε, αρκεί, αλλά θέλουμε να, παρόλα αυτά να κάνουμε πιο αποτελεσματικούς τους ελέγχους και πιστεύω ότι σημειώσαμε πρόοδο για να καταλήξουμε σε συνένεση επ' αυτού, κάτι που δείχνει ότι είναι κατάλληλοι αλλά και παρκώς ευέλικτοι κανόνες του Σέγγεν, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Έρχομαι τώρα στα εσωτερικά σύνορα και την κατάσταση εντός του χώρου του Σέγγεν. Δυστυχώς έχουμε να κοινώσουμε ότι δεν υπάρχει επαρκή πρόοδο ότι αφορά τη χαρτογράφηση της κατάσταση των δευτερογενών κινήσεων, δηλαδή ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής αλλά μπορούν να μετακινηθούν από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Μαζί με τον Frontex πριν από 2-3 χρόνια ε, συνεργαστήκαμε για να βρούμε ε, ή να κάνουμε αξιολόγηση και επισκόπηση τη κατάσταση, βασισμένη σε στοιχεία, πόσα κράτη-μέλη, πόσα άτομα. Κάποια κράτη όμω δεν έχουν δώσει ακόμα στη Frontex τα στοιχεία ώστε να έχουν μια συνολική εικόνα. Όπω πάντα, τρει υποθέσει κρατών μελών είχαμε που επανεισήγαγαν ελέγχου στα εσωτερικά του σύνορα για μια εβδομάδα, προσωρινά δηλαδή. Επίση, όπω και στο παρελθόν, η Κομισιόν δεν θεώρησε ότι υπάρχει λόγο να αμφισβητηθούν τα μέτρα αυτά ή οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτά. Ωστόσο, επισημαίνουμε στην έκθεση ότι δεν θεωρούμε εντελώς ικανοποιητική ε, την ε, υποβολή αναφορών ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη για το πώς αποτελεσματικά και αναλογικά ήταν αυτά τα μέτρα, πώς επηρέασαν την ελεύθερη κυκλοφορία κτλ. με βάση τα διάφορα κριτήρια που έχουμε στον κώδικα σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση του Σέγγεν. Την ώρα που μιλάμε λίγο πολύ, έληξε ο παλαιός μηχανισμός και άρχισε να ισχύει ο νέος. Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την πλήρη εφαρμογή του μηχανισμού αυτού το 2015 με την έγκριση όλων των λοιπόν παρασκευαστικών εγγράφων. Το 2015, στο πλαίσιο του τακτικού χρονοδιαγράμματος που έχουμε, θα αξιολογήσουμε το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία και το Λίχτενστάιν για όλους τους τομείς του κεκτημένου του Σέγγεν και επιπροσθέτως θα προβούμε και σε ε, μη ανακοινωθήσεις εκ των προτέρων επισκέψεις ε, σε κάποια χερσαία σύνορα. Επίσης με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρξε ακόμη απόφαση του Συμβουλίου για την άρση των ε, ελέγχων στα σύνορα με τη Ρουμανία και την Βουλγαρία. Ελπίζουμε να συμβεί όμως σύντομα αυτά. Τέλος, ό,τι αφορά τα συμπεράσματά μας, επισημαίνουμε στην έκθεση τρία ζητήματα για τα οποία χρειάζεται συζήτηση και θα θέλαμε να έχουμε και τις δικές σας απόψεις όπως και του Συμβουλίου. Πρώτον, ετοιμότητα στα ανατολικά σύνορα. Αν αλλάξει κατάσταση στο μέλλον, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή. Έχουν ε, λάβει ή μπορούν να λάβουν ε, τα κράτη-μέλη τα μέτρα, έχουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες μαζικές εισρωές. Δεύτερον, αναστευτικέ ροές. Υπάρχει κάτι στη διακυβέρνηση του Σέγγεν που μπορεί να βελτιωθεί ή χρειάζεται ίσως να αλλάξει λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τις μεταναστευτικές πιέσεις. Και υπάρχουν και άλλες πολιτικές που συνδέονται στενά, όπως είναι πολιτική ασύλου ή η συνεργασία με τρίτες χώρες. Και το τρίτο, πιο πρακτικό ζήτημα για το οποίο θα θέλαμε να έχουμε feedback από τα κράτη-μέλη, για τη χρήση ε, του συστήματος ενημέρωσης για τις θεωρήσεις. Ποια είναι η εμπειρία των κρατών μελών μέχρι τώρα. Εδώ ολοκληρώνω. Αλλά κύριε Πρόεδρε, είμαι έτοιμο να απαντήσω με τα χαρά στι ερωτήσει των συναδέλφων. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίλσεν. Σύντομη παρουσίαση, μεστή όμω. Και θέσατε και τρία μείζωνα ζητήματα και ερωτήματα. Πολύ σημαντικά, ιδίω αυτό το σύστημα πληροφοριών, θεωρήσεων, διαβατήριων και τα ανατολικά σύνορα. Δυστυχώ δεν είναι τόσοι πολλοί βουλευτέ ε, στην αίθουσα αλλά πολύ σημαντικά τα θέματα και πολύ σημαντικός και ο τομέας. Θα δώσω το λόγο σε έναν από τους ειδήμονες για το θέμα αυτό καταρχάς. Ο Κάρλος Κοέλιο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα ευχαριστούμε για αυτή την ε, τόσο λεπτομερή έκθεση που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά συντεταγμένη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Το ένα είναι οι αριθμοί τους οποίους παρουσίασε η Κομισιόν όσον αφορά την παρουσίαση των μεταναστευτικών ρευμάτων ε, και της, των, της απώλειας ανθρώπινης ζωής στη Μεσόγειο, αριθμοί που αυξάνονται δυστυχώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην Ιταλία, προς την Ιταλία και προς την Ελλάδα αυξάνονται τα μεταναστευτικά ρεύματα και αυξάνονται και, αυξάνεται και ο αριθμός των τον άσυλο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και αυτή τη διαπίστωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο μάλλον είναι κατάλληλα προ, ε, προσαρμοσμένο ε, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πρέπει απλώς να εφαρμοστούν οι ισχύοντες ε, κανόνες. Γι' αυτό το λέω, διότι υπάρχουν διάφορες... Ε, διάφορες απόψεις που ακούγονται, ίσως λαϊκιστών, που λένε ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Όχι, δεν πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες, πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες, σωστά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό για αυτή την τόσο λεπτομερή ανάλυση και η... γιατί ασχολήθηκε και με την επαναφορά των ελέγχων σε εξωτερικά σύνορα. Ε, Αυτός δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δίκιο όταν συμπεριέλαβε ε, κάποια κριτήρια για την εφαρμογή του νέου μηχανισμού. Σας υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο δεν συμφωνούσε απόλυτα με τις ε, απαιτήσεις μας αν θέλετε και ε, αυτό ε, το αποδεικνύει και η έκθεση της Κομισιόν. Υπάρχει, και θα ήθελα να ευχαριστήσω μάλλον την Κομισιόν για την πρότασή της και για την προσπάθεια προσπάθεια και την θέληση να υποστηρίξει τις χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα όλες τις οδηγίες ε, τον επόμενο Φεβρουάριο θα γίνει μια αναθεώρηση του συστήματος και μια ε, εκτίμηση της εφαρμογής του συστήματος. Υπάρχουν επίσης και οι μη προαναγγελθήσεις ε, επισκέψεις. Ε, αυτό είναι ένα, ε, ένα κείμενο το οποίο ήταν δύσκολο να γίνει δεκτό, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι μη προαναγγελθήσεις επισκέψεις είναι ζωτική σημασία για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά το σύστημα Schengen. Για το 6 ε, εδώ το κοινοβούλιο έχει δίκιο. Ο μηχανισμός που προβλέπετε εδώ είναι πολύ χρήσιμος, αλλά τα προβλήματα τα οποία είχαμε εντοπίσει τότε ήταν προβλήματα ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Κομισιό είχε ζητήσει στα κράτη-μέλη να καταβάλουν ε, περαιτέρω προσπάθειες στα θέματα της ασφάλειας. Ότι η, και ότι η έλεγχη αυτή δεν θα πρέπει να ε, δίδονται εργολαβικά σε εξωτερικές υπηρεσίες ε, πρέπει να ε, γίνονται από τις κρατικές, από τις εθνικές υπηρεσίες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Υπάρχει ένα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μιλάνε και ιδίω ε, για φύλακες των συνόρων που μιλάνε για ένα μεγάλο αριθμό λαθών που γίνονται κυρίως στα βιομετρικά στοιχεία και στα δακτυλικά αποτυπώματα. Γίνονται λάθη όταν συλλέγονται τα δακτυλικά αποτυπώματα και ε, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση γίνεται κάπως επικίνδυνη. Θα πρέπει επομένως να ασκηθεί κάποια πίεση έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα αυτών των στοιχείων. Ευχαριστώ. Okay, um, next speaker is, uh, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριο, η κυρία Ρεβέτα Πολυφάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ η έκθεση αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός ασυμβατότητας μεταξύ των ενεργειών των κρατών μελών και του κοινοτικού κεκτημένου, δηλαδή όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την διοικητική κράτηση και υπάρχουν, υπάρχει θέληση από πλευρά της Κομισιόν να ξεκινήσουν διαδικασίες κατά κάποιων χωρών. Ε, για παραβίαση υποχρεώσεων. Ε, σε τι, σε τι, πού ακριβώς θα στηριχτείτε, ας πούμε για τα κέντρα ε, κράτησης που χρησιμοποιούν πολλά κράτη-μέλη, η κράτηση είναι το τελευταίο ε, εργαλείο, όργανο που πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα κράτος μέλος. Κάποια, οι μετανάστες και τα παιδιά κυρίως κρατούνται σε μέρη τα οποία δεν είναι ε, κατάλληλα, πολλές φορές παραβιάζονται τα δικαιώματα των μεταναστών. Επίσης η Κομισιό ε, αναφέρεται και σε άλλα μέτρα πέραν της κράτησης. Ε, εσείς έχετε κάποια παραδείγματα να μας παρουσιάσετε. Παραδείγματα σε κάποια κράτη-μέλη. Κύριε Σεγκυριάνου, ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, το 3-6 της έκθεσης αφορά, όπου η Κομισιόν λέει ότι στηρίζει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την πρόσβασή τους στο χώρο Σέγγεν. Τι, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις εδώ. Μπορεί να μας ενημερώσει με κάποια καινούρια στοιχεία. Τώρα, το 4-3 της ίδιας έκθεσης αφορά την πολιτική των θεωρήσεων και συμφωνίες επανεισδοχής. Η Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Πολωνία, Ρουμανία έχουν στείλει ε, κοινοποίηση σε σχέση με καταστάσεις μια αμοιβαιότητας που αφορούν κάποιες τρίτες χώρες, ε, μεταξύ αυτών είπα και Αυστραλία. Η ερώτηση είναι, προβλέπει η Κομισιόν ε, περαιτέρω μέτρα, θα αναμένουμε νέες εξελίξεις ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπίργκιτ Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι βρίσκω τη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Συζητάμε για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακούμε προκειμένου περί συνοριακών ελέγχων ότι υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για το πώς θα διεξάγονται αλλά προφανώς δεν γίνονται παντού όπως πρέπει και τα κράτη-μέλη δεν διασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών κανόνων από τους τοπικούς αξιωματικούς και εργαζομένους. Εις ό,τι αφορά το χώρο Σέγγεν, πάλι φαίνεται ότι υπάρχουν αιτήματα σχετικά με το τι μπορεί να γίνει, αλλά σχετικά λίγο ε, αποτέλεσμα ε, επιτυγχάνουμε. Πού είναι τα κενά λοιπόν που πρέπει να κάνουμε κάτι ή πρέπει να επιβάλλουμε με τρόπο αποτελεσματικό τα υφιστάμενα μέτρα για, και στα εξωτερικά σύνορα. Ε, σε ό,τι αφορά το θέμα Ρουμανία, Βουλγαρία και προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν, αυτό είναι μια ατέρμονη ιστορία. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο νομίζω ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό και ο κύριος Νίσης από ό,τι κατάλαβα ελπίζει σύντομα να υπάρξει κάποια κίνηση σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν το βλέπω ακόμα. Ίσως όμως εσείς έχετε συγκεκριμένους λόγους για να είστε αισιόδοξο. Κύριε Νίλσεν, η σειρά σας και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Να αρχίσω από το τελευταίο. Δυστυχώς δεν προσπαθούσα να φανώ αισιόδοξο σχετικά με την Βουλγαρία-Ρουμανία. Ήθελα να είμαι ουδέτερος. Με βάση τις πληροφορίες που έχω εγώ, δεν έμεινε στην ε, ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ΔΕΗ την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν θα γίνει τίποτα από αυτής της Προεδρίας. Ελπίζουμε όμως ότι η επόμενη Προεδρία, το επόμενο εξάμεινο θα γίνουν ανανεωμένες προσπάθειες των κρατών μελών για εξέβρεση συμφωνίας. Τώρα για τις άλλες ερωτήσεις. Ε, θα πρέπει να ελέγξω κάποια στοιχεία και να επανέλθω. Ιδιαίτερα ίσως ό,τι αφορά την οδηγία για την επιστροφή πρέπει να δω αν έχουμε φτάσει στο σημείο που ελήφθη απόφαση σχετικά με το, τις ε, διαδικασίες ε, επί παραβάση που θα κινηθούν και κατά ποιών κρατών μελών. Για την κράτηση έχουμε κάνει κάποιες μελέτες κατά το παρελθόν και σε συνεργασία με τον οργανισμό ΦΡΑ για τα θεμελιώδη δικαιώματα που εντοπίζει βελτίστες πρακτικές και λέει και τα κρατη που έχουν τις καλές αυτές πρακτικές. Θα δούμε, θα, το δούμε και θα προωθήσουμε τις απαντήσεις. Για την αμοιβαιότητα στις θεωρήσεις συνεχίζεται ο διάλογος με τις σχετικές ε, τρίτες χώρες ε, και για τα, κράτη, τα πέντε κράτη-μέλη που έκαναν ανακοινώσεις. Επίσης, πράγματι είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ε, πληροφορίες επιτόπου αν δείτε το χώρο Σέγγεν και τα εξωτερικά σύνορα που είναι τόσο μεγάλα, ε, αντιλαμβάνεστε ότι καμιά φορά είναι δύσκολο να ξέρουμε σε καθημερινή βάση πώς εφαρμόζονται οι κανόνες από τα κράτη-μέλη. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος ε, μηχανισμός του Σέγγεν θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία, πιο συγκεκριμένα και σε συνεργασία με τους οργανισμούς μας, ε, Frontex και τον οργανισμό ΦΡΑ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, θα ε, έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε κλείνουμε τη συζήτηση αυτή. Ωραία, συναδελφοί. Το επόμενο θέμα μας είναι οι ψηφοφορίες που προβλέπονται όμως για τις 12 και 4. Αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. Θα ήθελα θα, να ψηφίσουμε τώρα, αλλά βλέπω πολλοί να διαφωνούν. Ναι. Υπάρχουν μερικοί που έχουν κάνει το λογαριασμό τους για να έρθουν και ακριβώς στις 12 και 4, οπότε υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ας κάνουμε διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα θα είναι αυτό. 12 και 14 να είστε όλοι εδώ, μην καθυστερήσουμε. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Για μένα θα μου άρεσε πολύ να ψηφίσουμε τώρα. Αλλά πώς θα γίνει. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε στις 12 και 4 γιατί άλλοι συνάδελφοι το γνωρίζουν αυτό και έχουν κάνει ε, το πρόγραμμά τους. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η σειρά για τις ψηφοφορίες. Ε, πρώτο θέμα, καταρχάς πριν πω ποιο είναι το θέμα, έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας. Και αν ναι, παρακαλώ να τις αγάγετε στο μηχάνημα και να καθίσετε για να μην καθυστερήσουμε. Μία ψηφοφορία έχουμε σήμερα. Για τη δεύτερη, το θέμα 10 αναβλήθηκε, δεν το ακούσατε όσοι δεν ήσασταν παρόντες. Θα ψηφίσουμε μόνο την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος για αυτή την στρατηγική εσωτερική ασφάλεια. 6 Οκτωβρίου αποφάσισαν να ε, καταθέσουν οι συντονιστές, να καταθέσουν μάλλον μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το θέμα. Προβλέπεται συζήτηση για το Δεκέμβριο. Αν εγκριθεί σήμερα αυτό ε, το ψήφισμα θα κατατεθεί στην Ολομέλεια ψήφισμα της ΛΥΠΕ για την ολοκλήρωση της συζήτησης και η Κομισιόν θα το λάβει υπόψη της για την εκπόνηση της νέας ε, Στρατική εσωτερικής ασφάλειας. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες για τη δουλειά τους και για τις κοινέ τους προσπάθειες ε, να βρούμε μια συμφωνία. Σας καλώ να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου. Παρακαλώ, έχετε ζήτημα επί της διαδικασίας. Ναι, θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες παρακαλώ. Να μας πείτε, λέει ο Πρόεδρος, ποια είναι η προφορική τροπολογία. Στην τυπολογική ε, σκέψη Β. Αύξηση των μεταναστευτικών ροών και ταχαίως αναπτυσσόμενος ε, ριζοσπαστισμός και εξτρεμισμός και ε, σχέση με μετανάστευση, θέματα ασφάλειας, το Ισλαμικό κράτος. Στο ΣΥ, στη τηλεοπτική σκέψη Γ για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία πλήρη στρατική εσωτερική ασφάλεια, αυτή θα πρέπει να σέβεται τι εθνικέ αρμοδιότητε σε κάποιου τόμει σα πολιτική ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των κρατών και προστέμενη αξία, ιδίω στον τομέα των εσωτερικών ελέγχων. Κώδικα θεωρήσεων Σέγγεν και ξένοι μαχητέ. Στο 4, στο άρθρο 4, μια προσθήκη ξένοι μαχητές και εγχώρια τρομοκρατία, διακίνηση ανθρώπων, εκμετάλλευση παιδιών. Στο 4α, αλλαγή. Αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενε στρατηγικές τη Ευρωπαϊκής στον τομέα αυτό έχουν αποτύχει και δεν αντιμετώπισαν τα ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας με ολιστικό τρόπο. Σε σχέση με τα προβλήματα της ασφάλεια σε περιοχές που γεννιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι οι στρατικές αυτές συνεισέφεραν ε, στο να δημιουργηθεί τελικά ένας φαύλος κύκλος, όπου άτομα από την Ένωση ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για να λάβουν μέρος σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και έχουν αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε κοινωνικό αποκλεισμό μεταξύ των κοινοτήτων των μεταναστών και επακόλουθο ήταν η ρισοσπαστικοποίηση ορισμένων. Αν δεν υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων φορέων, οι μελλοντικές στρατηγικές της Ένωσης ε, κινδυνεύουν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν αυτόν τον φαύλο κύκλο ή και να τον οξύνουν ακόμη περισσότερο. Άρθρο 5, αλλαγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει αύξηση της θρησκευτική μυσαλλοδοξίας στην Ένωση και στις γειτονικέ χώρες. Και η στρατολόγηση ξένων μαχητών είναι και η πλέον ε, ανησυχητική απειλή και εντός και εκτός Ένωσης. Καλεί λοιπόν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν κάθε δυνατή δράση για την μεγιστοποίηση ε, της χρήσης της ισχύουσας νομοθεσίας ε, για να αποτρέψουμε την αύξηση του εξτρεμισμού και αποκινούμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουμε σε συνεργασία και με τον ΟΗΕ νέα μέτρα για την πρόθεση της Παγκόσμια Ειρήνης και Ασφάλειας. Έχουμε και στην παράγραφο 9 μια προσθήκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αμβέμπιστοσύνη σύνυμα αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με σεβασμό της ε, πολυμορφίας των νομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγραφος 11. Παράγραφος 11 προσθήκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι αυτή η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη ε, στα μέσα και την ουσία, ώστε α, χώρες που απειλούνται με τις ίδιες έχουν τις ίδιες απειλές, θα πρέπει να καλούνται σε συζητήσεις για την εξέβαση κοινών λύσεων στα κοινά προβλήματα χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, ειρήνης και ασφάλειας ή πολίτες θα πρέπει να ε, δίνουν τη γνώμη του με βάση τι ανάγκε του τι καταστάσει που αντιμετωπίζουν ιδίω στον τομέα των συμφωνιών επανεισδοχή, δημιουργία υποδομών, ανταλλαγή πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι ο συντονισμός και η συνεργασία είναι ευεργετικός εάν γίνεται με ταυτόχρονα σεβασμό στι αρχές της ιδιοκτησίας και τη επικουρικότητα. Παράγραφό 13 πρέπει να διαγραφεί. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Um, Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον κανόνα με το, του καταστατικού, θα πρέπει να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για αυτές τις τροπο, ε, προφορικές τροπολογίες ε, κάθετος ομιλία που ακούσαμε. Λοιπόν, Υπάρχουν πάνω από τέσσερις αντιρρήσεις, επομένως σύμφωνα με το 169 δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις προφορικές τροπολογίες. Προχωράμε στην ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 30 υπέρ 4 κατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 38 υπέρ, 4 κατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, τελειώσαμε.